Mesdames, Messieurs, je vous Να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας ενημερώσω καταρχήν για τις αλλαγές που έχουν γίνει στις εργασίες μας. Έχει τροποποιηθεί και η ημερήσια διάταξη. Το σημείο 10 και το σημείο 15 αναβάλλονται. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις ε, για την ημερησία διάταξη και δεν βλέπω, θεωρείτε ότι εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να σας ενημερώσω ότι η συνεδρίαση μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Οπότε κατανοείτε ποιες είναι και οι συνέπειες. Όλοι αυτοί που ενδιαφέρονται για την συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, κρίνουν το έργο σας και τις ευθύνες σας. Δεν έχω άλλες ανακοινώσεις, επομένως ε, θα περάσουμε αμέσως ε, στα επόμενα σημεία της ημερησίας διάταξης, δηλαδή στις εργασίες που έγιναν από την κυρία Μωρίς Σαρτιέ και την κυρία Ζιεύσκα ό,τι αφορά τα δικαιώματα των παιδιών στις διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές. Πριν να μπούμε στη συζήτηση, θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη των Επιτροπών ΠΕΤ και ΦΑΜ που απάντησαν στην πρόσκλησή μας και φυσικά θα προσπαθήσω να τους δώσω το λόγο στις 2,5 ώρες. Η κυρία Μερασιαρτιά θα προεδρεύσει τη συζήτηση και αν χρειαστεί θα τη βοηθήσω κι εγώ. Όμως, ε, καθώς ε, είναι ειδική στο θέμα, καλό είναι να δώσετε εσείς το λόγο έτσι όπως ε, κρίνετε καλύτερο. Επομένως, έχετε το λόγο, αγαπητή Λιζαπέτ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Ζαν Και εγώ χαίρομαι πολύ που θα εγκαινιάσω αυτή την ακρόαση που αφορά τα δικαιώματα των παιδιών ε, στις διασυνοριακές οικογενειακές ε, διαφορές. Και πάλι χίλια ευχαριστώ στην Επιτροπή Νομικών ε, Υπόθεσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μας υποδέχεστε γιατί είναι πραγματικά μια ολόκληρη ομάδα που έχει κινητοποιηθεί για το θέμα των δικαιωμάτων των παιδιών. Επίσης, ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, Γιούρη για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε μεταξύ της Επιτροπής ε, και του δικού μου γραφείου, όχι μόνο για την οργάνωση της ακρόασης αυτής, αλλά και σε όλη την καθημερινή μου εργασία ως συντονίστρια για τα δικαιώματα των παιδιών θα ήθελα να πω και ε, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε συνάδελφο Ταντία Βιάσκα, καθώς ε, είναι η συγκήτρια για τον κανονισμό Βρυξέλλε 2, Βρυξέλλες 2α και θα δείτε πόσο έχουμε κινητοποιηθεί αγαπητοί συνάδελφοι και πόσο χρειάζεται να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ε, για να προωθήσουμε αυτή την προβληματική. Από το 1997 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε αναγνωρίσει τη σημασία του προβλήματος ε, των διασυνοριακών απαγωγών παιδιών, δημιουργώντας ε, το λειτουργήμα του διαμεσολαβητή. Μέσα σε 30 χρόνια πολλοί γονείς ζήτησαν τις δικές μας υπηρεσίες για να ε, μπορέσουν να αντιμετωπίσουν διάφορες νομικές ε, και ιδιαίτερα πολύπλοκες συναισθηματικά και επώδυνες καταστάσεις. Επώδυνες και πολύπλοκες για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς και φυσικά και για το σύνολο των οικογενειών. Τον Απρίλιο 2018 διευρύνθηκε ε, η εντολή μου για να αντικατοπτρίσω τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συνομοθέτη να εγγυηθεί για να προστατεύσει τα δικαιώματα των παιδιών ε, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό το νέο λειτουργήμα ονομάζεται Συντονίστρια για τα Δικαιώματα των Παιδιών επανεπιβεβαιώνει και καθιερώνει τη δέσμευση αυτή και με ιδιαίτερη υπερηφάνεια τον λαμβάνω. Από την έναρξη αυτής της εντολής ε, και ε, από τότε που αρχίσαμε να βοηθάμε τους γονείς, εγώ θέσπισα ε, ένα ολόκληρο προβληματισμό για τα δημιουργία των παιδιών στις συνορικές οικοκοινικές διαφορές και εξεπλάγει, καθώς διαπίστωσε ότι για κάθε μεμονωμένη περίπτωση τόσοι επαγγελματίε, τόσοι οργανισμοί και τόσα ιδρύματα μπλέκονται δικηγόροι, δικαστές, υπάλληλοι, κοινωνική λειτουργία, αστυνομική. Είναι μακροσκελής ο κατάλογος και πολλά άτομα είχα, έχουν την ευθύνη να προστατεύσουν και να εγγυηθούν τα δικαιώματα των παιδιών αυτών. Ξέρω για τις εμπειρίες, για τις πείρες μου, ότι όλοι οι επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα αυτό είναι άνθρωποι με μεγάλο πάθος και με δέσμευση, όμως δυστυχώς δεν είναι ιδανική η κατάσταση. Πολλά απομένουν να γίνουν για να προσαρμόσουμε τις νομικές και διοικητικές μας διαδικασίες στις ανάγκες και στα δικαιώματα των ενδιαφερομένων παιδιών. Καθώς κατά τη διάρκεια αυτών των οικογενειακών διαφορών υπάρχουν ακόμη πολλά παιδιά τα οποία τα αποστερούν με τη σχέση με τον ένα από τους γονείς τους και πολλές φορές αυτό συμβαίνει για μήνες, για χρόνια και μερικές φορές και για πάντα. Πού είναι λοιπόν η αρχή του ε, του συμφέροντος του παιδιού που τόσο συχνά αναφέρουμε και που θα πρέπει ε, εδώ ε, να τη λάβουμε υπόψη στα γεγονότα. Ήθελα να οργανώσω αυτή την ακρεώση γιατί είμαι επιβεβαισμένη ότι αυτό το θέμα είναι ζωτικό και πήγον. Αλλάζει ο κόσμος, ε, αυξάνεται ο αριθμός ε, των ε, διασυνοριακών οικογενειών ε, και έτσι πολλές φορές αυξάνονται και τα διαζύγια. Σήμερα χαίρομαι που θα ακούσουμε ένα πάνελ εμπειρογνωμόνων με διεθνή αναγνώριση θα δούμε ποιες είναι οι διάφορες δυνατότητες ανάληψης ε, δράσης και προβληματισμού. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίε και κύριοι για την παρουσία σας. Χαίρομαι που μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας τις ε, πλούσιες εμπειρίες σας και τις βέλτιστες πρακτικές που διέπουν την καθημερινή σας εργασία ως ε, δικαστές, αστυνομικοί διαμεσολαβητές, επαγγελματίες του δικαίου και την ε, ε, προηγούμενη της ε, ημέρας, της Παγκόσμιας ημέρας για τα δικαιώματα του παιδιού. Αυτή η διάσκεψη θα δηλώσει τη δέσμευσή μας να εργαστούμε μακροπρόθεσμα για να αγγιθούμε τα δικαιώματα των παιδιών για να έχουμε μια δικαιοσύνη πιο προσαρμοσμένη στις δικές τους ανάγκες. Θα δώσω το λόγο τώρα στο συνάδελφο Τέους Τζιέσκα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φίλο και εισηγητή για τον κανονισμό Βρυξέλλες 2α σε σχέση με την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων για γαμικές υποθέσεις και για την γονική ευθύνη. Έχετε το λόγο κύριε Βιέσκα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μωρή Σαρτιέ. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη σημερινή ακρόαση. Η ακρόαση αυτή αφορά σε ένα θέμα οικογενειακού δικαίου ιδιαίτερα σημαντικό και κυρίως σημαντικό γιατί ενδιαφέρει άμεσα τα παιδιά ιδιαίτερα στην περίπτωση σοβαρών οικογενειακών διαφορών σε περιπτώσεις ε, τέτοιου είδους ε, διαφορών ο πιο αδύναμος κρίκος είναι φυσικά το παιδί γιατί το παιδί πολύ συχνά δεν είναι σε θέση να κατανοήσει την περιπλοκότητα των προβλημάτων που έχει μπροστά του. Εδώ και αρκετό καιρό εγώ προσωπικά έχω ενδιαφερθεί και εργαστεί για το θέμα το συγκεκριμένο. Έχω μιλήσει με πολλούς εμπειρογνώμονες, Έχω μιλήσει με μέλη της νομικής κοινότητας, έχω μιλήσει με εμπειρογνώμονες εκτός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ασχολούνται με περιπτώσεις τέτοιου είδους που ενδιαφέρουν τα παιδιά. Και το μόνο συμπέρασμα στο οποίο μπόρεσα να καταλήξω είναι ότι τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε τους τελευταίους μήνες έχουν τη σωστή πορεία, ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό το οποίο είναι προβληματικό βέβαια είναι η ταχύτητα την οποία έχουμε, η οποία δυστυχώς είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου και της εργασίας μου στο Κοινοβούλιο κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η βιασύνη φυσικά δεν είναι κάτι το παραγωγικό. Πολλές φορές απαιτείται περισσότερος χρόνος που οδηγεί σε καλύτερες ρυθμίσεις. Αλλά για ένα θέμα τόσο σημαντικό όσο τα δικαιώματα των παιδιών, έχω την αίσθηση ότι τα θεσμικά όργανα, όπως επίσης και οι εκπρόσωποι των κρατών μελών, θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους ακόμα περισσότερο και να εμπλακούν ακόμα περισσότερο σε αυτού του είδους την προσπάθεια έτσι ώστε οι διαδικασίες αυτές οι εξελικτικές προς τη σωστή κατεύθυνση να επιταχυνθούν. Όλες οι αλλαγές αυτές φυσικά είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητες. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας μας μέχρι σήμερα, ιδιαίτερα για την αναθεώρηση των Βρυξελών 2α, στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Μόρα Σαρτιέ, είχαμε την δυνατότητα να οργανώσουμε πολλές συναντήσεις με εμπειρογνώμονες. Είχαμε την δυνατότητα να κάνουμε πολλές συζητήσεις με εκπροσώπους της νομικής κοινότητας και όλες οι συζητήσεις αυτές οδήγησαν, αν θέλετε, στο ίδιο συμπέρασμα. Ιεσδήποτε και αν είναι οι αλλαγές οι οποίες θα υπάρξουν στους κανονισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Αυτό το οποίο είναι σαφές ότι θα επηρεάσουν την ζωή των παιδιών και τα δικαιώματα των παιδιών και την ειδική θέση την οποία φυσικά έχουν ή πρέπει να έχουν τα παιδιά στις κοινωνίες μας. Αυτές λοιπόν οι αλλαγές θα πρέπει να είναι σε θέση ε, να αποδώσουν να ικανοποιήσουν τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει. Με άλλα λόγια η βασική μας ανησυχία είναι ε, φυσικά η ζωή των παιδιών μας. Όταν ασχοληθήκαμε με την αναθεώρηση της Σύμβασης Βρυξέλλες 2α, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αυτής και να συμπεριλάβει και το ε, θέμα της ε, γονεϊκής απαγωγής. Είναι κάτι το οποίο επιβαρύνει την οικογενειακή ζωή. Είναι κάτι το οποίο προκαλεί μεγάλη δυστυχία και στους γονείς αλλά και στα παιδιά. Και γι' αυτό λοιπόν προσπαθούμε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να ρυθμίσουμε το φαινόμενο αυτό συνειδητοποιούμε ότι ο αριθμός των μικτών ζευγαριών είναι κάτι το οποίο αυξάνεται συνεχώς και αυτό οδηγεί και στην αύξηση ε, των περιπτώσεων οικογενειακών διαφορών σε διαμεθοριακό επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε ακόμα περισσότερη προσοχή στο θέμα αυτό και να προσπαθήσουμε να δούμε ποια είναι η θέση ε, ενός παιδιού σε μια οικογένεια η οποία βρίσκεται στη διαδικασία αποσύνθεσης. Έχουμε καταλήξει μέχρι τώρα λοιπόν στο συμπέρασμα ότι στην περίπτωση κατά την οποία θα θέλαμε να δώσουμε στο παιδί τις δυνατότητες τις νομικές ε, τότε θα πρέπει να του προσδώσουμε τις ίδιες ευκαιρίες και δυνατότητες και τα ίδια δικαιώματα με έναν ενήλικο. Το παιδί πρέπει να έχει τα ίδια τουλάχιστον δικαιώματα και θα πρέπει να έχει φυσικά δικαίωμα επαρκούς εκπροσώπησης και μέσω των γονέων του ή και εκτός αν αυτό δεν είναι εφικτό. Συνεπώς η αναγνώριση των δικαιωμάτων των παιδιών πρέπει να είναι κάτι το υποχρεωτικό. Ακόμα και αν το παιδί έχει μια ηλικία κατά την οποία δεν είναι σε θέση να εκφραστεί, οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι τα παιδιά αυτά με μη προφορικό τρόπο έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας, έχουν την δυνατότητα έκφρασης. Είναι σημαντικό επίσης οι διαδικασίες εξέτασης των παιδιών να είναι σύντομες, να μην είναι περίπλοκες και να μην δημιουργούν τραύματα. Το παιδί θα πρέπει να τοποθετείτε σε μια οικογένειακή δαιμόνα ή σε, ένα ειδικό, ε, σε μια ειδική μονάδα φροντίδας να είναι σε θέση να ακούει και να εκφράζεται στην γλώσσα του και φυσικά υπάρχει και το μέσο της διαιτησίας. Η διαιτησία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον περιορισμό των αρνητικών συνεπειών τέτοιου είδους διαδικασιών. Ένα παιδί σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως όμοιρος σε οικογενειακές διαφορές ενηλίκων. Το ίδιο ισχύει και για τις υιοθεσίε σε διεθνές επίπεδο. Ο υπέρτατος λοιπόν στόχος, το υπέρτατο αγαθό το οποίο επιδιώκουμε είναι η ευημερία του παιδιού. Και εφόσον θέλουμε να προστατεύσουμε την ευημερία του παιδιού πρέπει να αυξήσουμε ταχύτητα. Θα ακούσουμε και τις απόψεις, τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Εμείς θεωρούμε, έχουμε δώσει προτεραιότητα στη διαδικασία αυτή. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε και να πετύχουμε. Θα ήθελα να δώσω τώρα τα μέλη του πάνελ στους τέσσερις εμπειρογνώμονες να προετοιμαστούν την δόκτωρα Άστριν Ποτζιαλότσκι, που μπορεί να πάρει το λόγο στην αίθουσα, την κυρία Χάτσινσον, τον κύριο Φρέντινγκ και τον Ανδρέα Σούλτς. Οκτώ λεπτά ο καθένας από εσά έτσι ώστε να υπάρξουν δυνατότητες απαντήσεων και στις ερωτήσεις οι οποίες ελπίζω ε, να εμπλουτιστούν μετά από την πρώτη σας παρουσίαση. Δόκτωρ Ποτζιαλόφσκι λοιπόν. Ξεκινάμε, είναι η πρώτη εμπειρογνώμων, είναι υπεύθυνη για τη Μονάδα Δικαιωμάτων των Παιδιών στην Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Δικαιώματα των Παιδιών και Δικαιοσύνη. Είστε ψυχολόγος, κοινωνική ψυχολόγος ε, και ασχολείστε με πολιτιστικά θέματα. Έχετε το λόγο για 8 λεπτά κυρία Ποτζιαλόσκη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. 8 λεπτά είναι λίγα, αλλά σε κάθε περίπτωση έχω και διαφάνειες τις οποίες θα διανέμω στη συνέχεια για να έχετε περισσότερες πληροφορίες. Τι γνωρίζουμε λοιπόν, με βάση μια εκτίμωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2,5 εκατομμύρια παιδιά εμπλέκονται σε δικαστικές υποθέσεις και ενώ ετησίως και παρότι υπάρχουν κάποια διεθνή πρότυπα θα πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες που είναι φιλικές προς το παιδιά, ειδικότερα όταν έχουμε περιπτώσεις ε, σοβαρής, ε, δηλαδή σοβαρές περιπτώσεις κυδαιμονίας ή περιπτώσεις απαγωγής ε, και παρόμοιες κατακράτησης. Και θα σας παρουσιάσω κάποια από τα βασικά. Τα καθήκοντα της δικής μας υπηρεσίας βασίζονται φυσικά στο άρθρο 12 της συνδίκης για τα θεμελιώδη δικαιώματα της των Ηνωμένων Εθνών και ε, έχουμε και το άρθρο 24 της, ε, του χάρτη κατά θεμελιώδη δικαιώματα με βάση το οποίο τα ε, τέκνα θα πρέπει να εκφράζονται ελευθέρωση και να βάνεται υπόψη η οριμότητα, ο βαθμό οριμότητά του. Και από εκεί και μετά υπάρχουν και κάποιε κατευθυντήρε γραμμέ, οι οποίε ορίζουν το πώ ακριβώ θα πρέπει να διαμορφώνονται αυτέ οι δικαστικέ διαδικασίε, έτσι ώστε τα παιδιά να νιώθουν άνετα. Ε, οι κατευθυντήρε γραμμέ τώρα του Συμβουλίου τη Ευρώπη ε, προβλέπουν κάποιε βασικέ αρχέ τη ε, μη διακριτική μεταχείριση, του βέλτιστου συμφέροντο του παιδιού, του να λαμβάνεται δεόντω υπόψη άποψη του παιδιού και η διεξαγωγή όλων αυτών των διαδικασιών με, μια, με έναν τρόπο και μια γλώσσα προσιτή φιλική προς το παιδί. Επίσης αναφέρεται το δικαίωμα πληροφόρησης του παιδιού και το δικαίωμα προστασίας το οποίο θα πρέπει να διασφαλίσετε. Και εδώ ε, μπαίνει και υψηλά ο πύχη σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των επαγγελματιών οι οποίοι ακριβώ έρχονται ε, σε επαφή με το παιδί. Άρα λοιπόν με βάση την έρευνα που εμεί ε, κάναμε εξετάσαμε ακριβώ την κατάσταση πολύ συγκεκριμένα και μπορούμε να περάσουμε εδώ στην επόμενη διαφάνεια Είδαμε λοιπόν ποια ήταν η εμπειρία 300 ε, ε, παιδιών από 10 διαφορετικά κράτη-μέλη και επίσης ζητήσαμε την άποψη δικαστών, ε, κοινωνικών λειτουργών, νομικών και ούτω καθεξής. Και ποια είναι τα βασικά πορίσματα με βάση τις εργασίες μας. Υπάρχουν πολύ διαφορετικές πρακτικές μεταξύ των διαφορετικών κρατών μελών αλλά και εντό των ίδιων κρατών μελών και εξαρτώνται αυτέ τι διαφορετικέ πρακτικέ συχνά από την κρίση του εκάστοτε επαγγελματία. Άρα λοιπόν ε, θεωρούμε πω θα πρέπει να υπάρξουν ενιαίε διαδικασίε έτσι ώστε για κάθε παιδί, ανεξαρτήτω τη κατάσταση που αντιμετωπίζει σε κάθε κράτο μέλο, να διασφαλίζεται ότι υπάρχει το δικαίωμα ακρόαση του, μπορεί να εκφράσει την άποψή του, έχει το δικαίωμα δηλαδή έκφρασή του και ε, μπορεί να το κάνει σε ένα ασφαλέ ε, περιβάλλον. Και επίσης όλα τα παιδιά τα οποία, των οποίων πήραμε συνέντευξη ανέφεραν ότι θέλουν να λαμβάνονται υπόψη, δηλαδή να γίνει ακρόαση και να έρθουν σε επαφή με εκείνον που είναι αρμόδιο τελικά για να τα λάβει τη σχετική απόφαση, αλλά χρειάζονται και την κατάλληλη πληροφόρηση πρωτού το κάνουν αυτό. Επίσης ε, χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα σε ό,τι αφορά το δικαίωμα ενημέρωση του παιδιού, δηλαδή να αναγνωρίζει ε, τι ακριβώ ε, συμβαίνει και να προστατευτεί, για παράδειγμα, το παιδί από διαδίκου του οποίου δεν θέλει να συναντήσει. Τέτοιου είδου δηλαδή διαδικασίε, τέτοιου είδου μέτρα δεν προβλέπονται, δεν αποτελούν συνήθη πρακτική στα κράτη-μέλη. Άρα λοιπόν ένα βασικό πόρισμα το οποίο πραγματικά επιβεβαιώθηκε από τη συνέντευξη με τα παιδιά, είναι επαγγελματική συμπεριφορά. Δηλαδή, αν επαγγελματία είναι εμ, εκπαιδευμένοι, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακριβώ και το κάνουν, να χρησιμοποιούν δηλαδή φιλική προ τα παιδιά ε, ε γλώσσα. Ε, και επίση ε, όταν έχουμε πολλαπλές ε, ακροάσεις ε, και τη σχετική ορολογία βέβαια τέτοιου είδους διαδικασίε είναι πολύ απειλητικές για τα κράτη-μέλη και μπορούν τέτοιου είδου διαδικασίε να καταστούν ακόμα πιο περιπλοκές. Οπότε εδώ υπάρχουν συγκεκριμένε κατευθυντήρε γραμμέ σε ό,τι αφορά τι τυποποιημένε πρακτικέ που θα πρέπει να ισχύουν. Επίσης θα ήθελα να τονίσω την σημασία του δικαιώματο ενημέρωση του παιδιού, δηλαδή του να γνωρίζει ακριβώ το τι συμβαίνει, ποια είναι η διαδικασία και να μπορεί να εκφράσει τη δική του γνώμη και θα πρέπει γι' αυτό το λόγο να υπάρχουν συγκεκριμένε διαδικαστικέ δικλείδε ασφαλεία. Για παράδειγμα, αν υπάρχει μια μαγνητοσκόπηση ε, μια ε, ακρόαση, ε, το παιδί φοβάται όταν δεν γνωρίζει τον λόγο, όταν γνωρίζει για παράδειγμα ε, ότι αυτό γίνεται για να μειωθεί ο αριθμό των ακροάσεων, ε, καθυσυχάζεται. Οπότε θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις εκείνε όπου το παιδί ακριβώ τα κατέχεται από φόβο και δεν μπορεί να συμμετάσχει κανονικά σε μια διαδικασία. Εάν δεν φοβάται, νιώθει άνετα το παιδί, μπορεί να κάνει και σαφείς τοποθετήσει, να, να, εκφράσει σαφώ τη γνώμη του. Και επίση θα πρέπει να λαμβάνονται και άλλα θέματα, όπω, για παράδειγμα, εάν θα πρέπει με το διάδικο να βρίσκεται στην ίδια αίθουσα ή όχι το παιδί ε, και ούτω καθεξής. Υπάρχουν δηλαδή διαδικασίες οι οποίες θα πρέπει να διασφαλιστούν προκειμένου ακριβώς η ενημέρωση που είναι κλειδί για το ε, παιδί μέσα σε μια διαδικασία να διασφαλιστεί. Ε, υπάρχουν ε, μία σειρά από διαφάνειε που έχω προετοιμάσει σε αυτή την παρουσίαση, αλλά υπάρχει και φυσικά η ίδια έκθεση. Υπάρχουν πολλές πρακτικές οι οποίες ανταλλάσσονται και στι οποίε μπορεί να αναφερθεί κανεί. και επίσης έχουμε ε, για το ζήτημα αυτό, ή την έννοια της αξιολόγησης της βαθμού οριμότητας του παιδιού. Εδώ δηλαδή τα σχετικά κριτήρια που αξιοποιούνται δεν είναι πολύ σαφή. Ε, δεν ε, υπάρχει σαφήνεια ως προς το πώς λαμβάνεται πώς υπόψη αυτός, αυτή η οριμότητα μέσα στην νομοθεσία και δεν γνωρίζουμε να λαμβάνει η χώρα συστηματικά μια τέτοια αξιολόγηση και μάλιστα η αναφορά αυτής της οριμότητας γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Άρα λοιπόν ο ίδιος τρόπος με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού είναι ο ίδιος με εκείνο της αξιολόγησης του βαθμού ρημότητας, δηλαδή πολύ διαφορετικό διαφορετικός κράτη-μέλη. Επίσης σε ό,τι αφορά το δικαίωμα προστασίας, θέλουν για παράδειγμα τα κράτη-μέλη να βρίσκονται μόνα τους σε μια αίθουσα με τον επαγγελματία ε, νομικό σε μια αίθουσα ή θέλουν για παράδειγμα να υπάρχει μια συνόδευση, να, να συνοδεύονται ε, καταφθάνοντας στην, ε, στην αίθουσα, να μην συναντήσουν ενδεχομένως τους γονείς. Ε, χρειάζονται λοιπόν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη και γι' αυτό στο πλαίσιο ακριβώς αυτού του δικαιώματος σε προστασίας ε, και υποστήριξης θα πρέπει να υπάρχει ένα αρμόδιο υποστήριξη στο παιδιό, ο οποίο, ε, οποίος συνοδεύει το παιδί καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδικασία και είναι ανεξάρτητο από του γονεί, γιατί συχνά αντιλαμβανόμαστε ή μάλλον αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα όπου θέτουμε πάρα πολλέ τέτοιε ευθύνε στου γονεί, οι οποίοι όμω δεν είναι αμερόληπτοι. Άρα λοιπόν η ύπαρξη ενό τέτοιου αρμοδίου θα μπορούσε να βοηθήσει ε, πολύ για την αντιμετώπιση αυτών των ε, μεροληπτικών τοποθετήσεων. Μένουν ε, μόλι 30 δευτερόλεπτα, οπότε ε, στο πλαίσιο του συμφέροντο ε, του παιδιού να αναφέρω ότι ε, θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία η οποία λαμβάνει υπόψη του διαφορετικού τομεί, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ακριβώ τη σαφή κατανόηση τη διαδικασία από το παιδί και υπάρχει και μια checklist που έχουμε προετοιμάσει για του επαγγελματίε από το χώρο σε ό,τι αφορά ακριβώ αυτά τα δικαιώματα του παιδιού σε ό,τι αφορά και μάλιστα διαφορετικότητα διαδικασίε ε, δικαστικέ ε, για διαφορετικέ υποθέσει και επίση έχουμε προετοιμάσει υλικό προκειμένου τα ίδια τα παιδιά να ενημερώνονται προ το ποια είναι τα δικαιώματά του, τι μπορούν να ζητήσουν. Ε, γιατί όταν το γνωρίζουν μπορούν ακριβώ να θέσουν τα δικά του ερωτήματα και να υποβάλουν τα δικά του αιτήματα. Κάτι τέτοιο κάνει τα παιδιά να ανέχουν πολύ πιο άνετα σε πλαίσιο μια διαδικασίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ε, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούσαμε και σας ευχαριστούμε που σεβαστήκατε και το χρόνο. Τώρα έχουμε την ε, κυρία Χάτσινσον. Είστε ειδική νομικός ε, σε θέματα οικογενειακών υποθέσεων στο Διεθνές Δίκαιο και στο Βρετανικό Δίκαιο επίσης είστε αρμόδια στο δικηγορικό γραφείο Dorson Κόνουελ στο Ηνωμένο Βασίλειο για θέματα που αφορούν τα παιδιά και έχετε και ειδική αναγνωρισμένη εμπειρογνωμοσύνη σε ό,τι αφορά τις διασυνοριακές διαφορές, σε ό,τι αφορά ε, την κυδαιμονία και τις απαγωγές παιδιών ε, δυνάμει και του κανονισμού Βρυξέλλες 2α ή της Σύμβασης της Χάγης. σας δίνω το λόγο και σας ευχαριστώ που ήρθατε για να καταθέσετε τις σκέψεις στη συζήτησή μας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα προσπαθήσω να σεβαστώ τα 8 λεπτά. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη του στην αίθουσα αν επανέλθω σε ένα-δύο βασικά, αλλά θα ήθελα καταρχήν ε, να ε, δούμε κάποιες διεθνείς συμβάσεις ε, που έχουν να κάνουν με την μετακίνηση των παιδιών και να δούμε πώς ε, σε μια χρονική περίοδο που έχει εξελιχθεί το δίκαιο στα κράτη-μέλη έχουμε ερμηνεύσει το νόμο μέσα από τα μάτια ε, του παιδιού και επίσης ε, μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους κινδύνους που μπορεί να θέτει αυτό για ένα παιδί. Έτσι λοιπόν τα παιδιά μετακινούνται στα διεθνή σύνορα για πολλούς λόγους, οι οικογένειες ε, μετακινούνται, δικαιούνται να μετακινούνται καθώς η ζωή μας γίνεται όλο ένα και πιο πολύπλοκη θα πρέπει λοιπόν να προβλέψουμε μηχανισμούς ε, για να αντιμετωπίσουμε ε, την ε, παράνομη μετακίνηση των παιδιών, όμως να μην δημιουργήσουμε ταυτόχρονα εμπόδια που να εμποδίζουν την νόμιμη μετακίνηση των παιδιών. Τι χρειάζεται όμως στις διεθνείς μας συμβάσεις είναι ασφάλεια σε επίπεδο πολιτικής αλλά και σε πρακτικό επίπεδο και καθώς ε, έχουν γίνει όλα ένα και πιο δύσκολες και πολύπλοκες ε, οι ζωές μας, γιατί όσοι εργάζονται στον κλάδο όλοι θα συμφωνούσαν ότι σε πάρα πολλές ε, περιπτώσεις απαγωγές παιδιών δεν μπορούμε να τις ταυτοποιήσουμε όλες αυτές τις περιπτώσεις Πολλές φορές είναι πολύπλοκες οι οικογένειες, μπορεί να να έχουμε τεροθαλή αδέλφια, και όπως είπα τα παιδιά μετακινούνται για πολλούς ε, λόγους και μερικές ε, φορές μπορεί να είναι για χρονικές ε, περιόδους που μπορεί να είναι μεγάλες αλλά όχι σε μόνιμη βάση. Και εδώ πρέπει να δούμε ποια είναι η νομολογία των συμβάσεων. Βλέπουμε λοιπόν την σύμβαση του 80 για τις αποδοχές των παιδιών και τη σύμβαση του 96 για την προστασία των παιδιών. Και βλέπετε εδώ στη διαφάνεια τις δύο αυτές ε, συμβάσεις. Έχουμε τη δομή και το πλαίσιο, απλώς θα πρέπει να δούμε τις αρχές δικαίου που θα πρέπει να ισχύουν και ποιο είναι το κράτος του οποίου το δίκαιο θα πρέπει να ισχύει για τα παιδιά και να διασφαλίσουμε ότι οι κανόνες ε, του ΟΗΕ ε, ισχύουν. Έτσι λοιπόν, Ας ε, φτάσουμε στο άρθρο 3 της ε, Σύμβασης του 1980 και της ε, υποκείμενη αρχή σε όλες τις καταστάσεις έχει να κάνει με την μετακίνηση ή την κράτηση του παιδιού παράνομα. Δηλαδή τα παιδιά μπορεί να μετακινούνται ή να κρατούνται σε ένα άλλο κράτος παράνομα και εφαρμόζοντας τη σύμβαση θα πρέπει να εντοπίσεις ποιο είναι το κράτος της συνήθους διαμονής του παιδιού τη στιγμή της ε, μετακίνησής του ή της ε, κράτησής του. Και ε, φυσικά εδώ οπωσδήποτε θα πρέπει να εφαρμοστεί η σύμβαση του 1980 αλλά και η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Αλλά ε, εκτός και αν μπορείς να δείξεις ότι ένα παιδί ε, ουσιαστικά μετακινήθηκε από ε, την ε, τοποθεσία της συνήθους ε, κατοικίας τότε θα πρέπει και να εφαρμοστεί και ο κανονισμός αλλά και η Σύμβαση των 96 όμως σε κανένα από αυτά δεν ορίζεται τι σημαίνει συνήθις κατοικία. Δηλαδή δεν ορίζεται που είναι η χώρα της συνήθους διαμονής του παιδιού. Και ε, ο ορισμός έχει εξελιχθεί μεταξύ των ε, διάφορων κρατών. Και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι βάσει της Σύμβασης της Χάγης δεν υπάρχει ε, κάποιο δικαστήριο ή νόμος που υπερισχύει. Κάθε κράτος εφαρμόζει τις δικές του χώρες διαδικασίες. Έτσι λοιπόν, αν δούμε τις εξελίξεις εντός ε, της Ευρώπης για το πώς προσδιορίζουμε την συνήθη κατοικία, η νομολογία είναι πάνω κάτω η ίδια στα κράτη της Δυτικής Ευρώπης για το πώς η εστίαση δίνεται στο παιδί για να προσδιορίσουμε την συνήθη κατοικία του παιδιού. δηλαδή, δεν ε, βλέπουμε απαραίτητα την πρόθεση των γονιών, ούτε τις συμφωνίες που έχουν γίνει ε, κάποια στιγμή, αλλά κοιτάζεις ε, το παιδί και κάνεις μια σειρά τεστ ε, για να δεις ε, το θέμα της σταθερότητας του παιδιού, το ε, βαθμό ένταξης που έχει πετύχει το παιδί για το αν ένα παιδί έχει δημιουργήσει κάποιες ρίζες και πώς έχει γίνει αυτό. Δηλαδή, το χάρη κάποια νεαρά παιδιά μπορεί πολύ γρήγορα να δημιουργήσουν αυτές τις ρίζες, ενώ άλλα παιδιά να χρειαστούν περισσότερο χρόνο. Όμως ε, αυτό δεν προσδορίζει απαραίτητα τη συνήθη κατοικία. Αν ένα ζευγάρι, παραδείγματο χάρη, πει ο άνδρα ε, έχω τώρα μία δουλειά και θα μετακομίσουμε από την Γαλλία στη Γερμανία για ένα χρόνο και μετακομίζει η οικογένεια μέσα σε αυτό το χρόνο. Σίγουρα δεν ήταν κάτι μόνιμο, όλοι τελικά θεωρούσαν ότι θα επιστρέψουν μετά από το ένα έτος, αλλά τώρα η εφαρμοστέα νομολογία στην Ευρώπη ε, μπορεί παραδείγματο χάρη μέσα σε αυτό το χρόνο τα παιδιά να έχουν χάσει τη συνήθι του κατοικία ε, στην ε, Γαλλία και να απέκτησαν καινούργια στη Γερμανία. Έτσι λοιπόν όταν τελειώσει αυτή η περίοδος, δηλαδή λέγει η σύζυγος όχι μου αρέσει το Βερολίνο και δεν θέλω να φύγω, ε, πάνε καλά τα παιδιά στο σχολείο, έχω γνωρίσει κάποιον άλλο κτλ. Μπορεί λοιπόν να ισχύει ότι ε, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει παράνομη κράτηση των παιδιών, γιατί ε, τη στιγμή που κρατήθηκαν τα παιδιά στη Γερμανία απέκτησαν τη συνήθεια κατοικία. Και θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό με τα δικαιώματα των παιδιών. Αυτό που θέλω να τονίσω εδώ στην ακρόση είναι το εξής ότι μία ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση ε, των απόψεων των παιδιών θέτει το παιδί σε κεντρικό ε, στάδιο. Δηλαδή, πέρα από το να δούμε τις αντιρρήσεις ε, των παιδιών, ε, εδώ θέτουμε το παιδί και τον προσδιορισμό του τι συμβαίνει στο παιδί στο κέντρο, στο επίκεντρο. Και αφού το κάνουμε αυτό, αν το κάνουμε αυτό, πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι για το παιδί, ποιες, πρέπει να παίρνουμε κάποιες να ακολουθήσουμε κάποιες διαδικασίες για να προστατεύσουμε το παιδί και να ακούσουμε τις απόψεις του παιδιού στη διαδικασία. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα πρακτικό ε, παράδειγμα ε, μία μητέρα με τα τέσσερα παιδιά της μετακόμισε στην Ισπανία. Ήταν νόμιμη η μετακίνηση αυτή, είχαν χωρίσει οι γονείς, συμφώνησε ο σύζυγος ε, και μετακόμισαν το καλοκαίρι. Τέσσερις μήνες αργότερα επέστρεψαν τα παιδιά στην Αγγλία για να επισκεφθούν ε, τον πατέρα για τις διακοπές των Χριστουγέννων ε, και στο τέλος των διακοπών τα κράτησε στην Αγγλία και είπε ότι δεν ήταν παράνομο αυτό γιατί ε, παρά το γεγονός ότι τα παιδιά είχαν πάει στην Ισπανία να ζήσουν με τη συγκατάθεσή του τα παιδιά στα εντετράμενη περίοδο δεν απέκτησαν συνήθεια κατοικία στην Ισπανία γιατί δεν είχαν εγκατασταθεί καλά ε, και ε, δεν τα πήγαιναν καλά στο σχολείο και το ανώτατο δικαστήριο ερευνώντας ε, από τα μάτια, από τη σκοπιά του παιδιού, το θέμα της συνήθους κατοικία, θεώρησε ότι δεν είχαν αποκτήσει συνήθη κατοικία <clears throat> και επομένως δεν ήταν άδικη η κράτησή τους, ε, δεν ήταν παράνομη η κράτησή τους στην Αγγλία. Έτσι λοιπόν ε, σας ζητώ να δούμε το θέμα της συνήθους κατοικίας υπό αυτό το πρίσμα όταν μιλάμε για την προστασία του παιδιού. Σας ευχαριστώ εκτιμήσαμε ιδιαίτερα το ότι χρησιμοποίησατε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δείξατε πού ε, δράζονται οι αρχές τις οποίες ακολουθείτε και αυτό διευκόλυσε και εμάς την κατανόηση του θέματος. Θα περάσω τώρα το λόγο στον κύριο Σίφερντινγκ. Ζητώ συγγνώμη αλλά δεν λέω το όνομά σας σωστά είσαστε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και γραμματέας της Νέστα, οικογένειας ΛΟΑΤ. Μία από τις αποστολές του δικτύου αυτού είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών που μεγαλώνουν σε οικογένειες αυτής της πολλαπλότητας έτσι ώστε να έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τα υπόλοιπα παιδιά προωθώντας πολιτικές εναντίον των διακρίσεων και ισότητας ευκαιριών. Σας ευχαριστώ για την εισαγωγή σας και την πρόσκλησή σας. Να σας μιλήσω εξ ονόματος του δικτύου μας λοιπόν. Ας περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Η ΝΕΛΦΑ είναι η ένωσή μας. Να πω ότι στις οικογένειες ουρανίου τόξου, όπως λέμε, υπάρχουν διακρίσεις εις βάρος των παιδιών, υπάρχουν ελλείψεις σε επίπεδο δικαιωμάτων και αυτό δημιουργεί δυσάρρωστες καταστάσεις ε, όταν ε, τίθενται θέματα ελευθερής διακίνησης παιδιών ή οικογενειών. Στο παρελθόν οι περιπτώσεις ήταν πολύ περίπλοκες σε περιπτώσεις διαζυγίου και απομάκρυνσης υπήρχε μια συνεχής ε, αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των παιδιών αυτών. Εδώ βλέπουμε ένα χάρτη. Ο χάρτης ε, του ουρανίου τόξου της Ευρώπης όπως λέμε. Εδώ υπάρχουν αναφορές στους νόμους και στις πολιτικές ε, οι οποίες αφορούν στους, στις κοινότητες ΛΟΑΤ σε σχέση με τα οικογενειακά δικαιώματα. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στη Δυτική Ευρώπη και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη με κάποιες εξαιρέσεις. Βλέπουμε τις δύο τελευταίες δεκαετίες, έχουμε πετύχει πολλά. Έχουμε ισότητα στον τομέα τον γαμικό. Έχουμε επίσης τις νέες δυνατότητες καταγραφής ε, των σχέσεων. Υπάρχουν έξι χώρες βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ε, δικαίωμα αναγνώρισης των ενώσεων αυτών. Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία, σοβακία Λετωνία και Λιθουανία. Αυτό επηρεάζει φυσικά τα παιδιά δεν θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα σε αυτό. Να πω ότι όταν υπάρχει ένας πατέρας ή μητέρα που δεν έχουν αναγνωριστεί νομικά, όταν δεν αναγνωρίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους, τότε μειώνονται οι αντίστοιχες δυνατότητες των γονιών, δημιουργούνται καταστάσεις αρνητικές για τους γονείς και φυσικά μείωση των δικαιωμάτων των ίδιων των παιδιών. Φυσικά η ελεύθερη διακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών και οι πολίτες και οι οικογένειές τους έχουν την δυνατότητα να κινούνται ελευθέρως, αλλά σε σχέση με τους ΛΟΑΤ τι μπορεί να σημαίνει κάτι τέτοιο. Πρόκειται για μια κανονική εταιρική σχέση, ε, τι γίνεται με, τα, με τις ενδιάμεσες κατηγορίες, ε, τι γίνεται με τα βιολογικά παιδιά, τι γίνεται με τα παιδιά δύο μητέρων. Υπάρχουν μερικές φορές κάποιες διευκρινήσεις στην λεγόμενη υπόθεση Κόμαν τον Ιούνιο. Υπήρξε μια απόφαση του Λουξεμβούργιου Δικαστηρίου και τώρα υπάρχει μια πρώτη αναγνώριση ε, για δύο γονείς δύο φίλου πλέον θα ήθελα να σας δείξω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να ζει κανείς ε, ε, σε μια τέτοια οικογένεια. Αυτή είναι η Φραντσέσκα, μια νεαρά κυρία που γεννήθηκε με σύστημα μηχανικής ανυπαραγωγής. Η μητέρα της είναι η Ελένη από την Ελλάδα και η κατοικία τους ε, είναι στην Ισπανία μητέρα, ε, η άλλη μητέρα είναι η Κέιτ. Το πιστοποιητικό γεννήσεως αναγνωρίζει και τις δύο μητέρες, ακόμα και χωρίς ε, να υπάρχει αναγνωρισμένος γάμος, αλλά πρέπει να καταγραφεί στο ε, ληξιαρχείο και του εξωτερικού οι χώρες όμως προέλευσης δεν δέχτηκαν η Ιταλία και η Ελλάδα. Η Ελλάδα είπε ότι δεν είναι δυνατό να υπάρξει καταγραφή στο ληξιαρχείο το ελληνικό γιατί δεν είναι εφικτό σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία να υπάρχουν δύο μητέρες και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην χώρα προέλευσης της άλλης μητέρας, υπάρχουν περιπτώσεις κοινή μητρότητας όπως λέγεται κάτω από ορισμένε προϋποθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι με κάποιες προϋποθέσεις. Μία προϋπόθεση είναι οι ε, θεραπείες γονιμότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κάτι το οποίο όμως δεν είχε κάνει η Κέιτ, οπότε ε, έμεινε άπατρης, δεν μπορούσε να πάρει διαβατήριο. Ε, στην Ισπανία διαγνώστηκε και με καρκίνο και έκανε ό,τι μπορούσε η οικογένεια για να αντιμετωπιστεί η ασθένεια του παιδιού, αλλά δυστυχώς δεν ήταν δυνατόν ε, να ταξιδεύει. Και στο τέλος ε, τελικά υπήρξε μια θετική κατάληξη, γιατί ένας δημόσιος υπάλληλος που ήταν υπεύθυνος για την καταγραφή ε, στην Ελλάδα του ληξιαρχείου, στο, στο Μητρό, έκανε τα στραβά μάτια. Και έτσι ε, μπόρεσαν να περάσουν στην απόκτηση της ισπανικής ε, ε, υπηκότητας, αλλά η Φραντσέσκα έτσι λόγω αυτής της κομπίνας εισαγωγικά έχασε τη μία μητέρα της τυπικά. Το επόμενο παράδειγμα έχει σχέση με αυτό που συζητάμε σήμερα. Είναι η ιστορία του Βικτόρ, αλλάζουμε φυσικά ε, τα ονόματα. Η μία μητέρα είναι η Τζάνετ από τη Δανία και η άλλη από την Βουλγαρία. Γεννήθηκε ο Βίκτος το 16 στην Δανία με κοινό πιστοποιητικό γέννησης και από τις δύο μητέρες, αλλά μετά από κάποιους μήνες χώρισαν και η μητέρα από τη Βουλγαρία προσπάθησε να πάρει ένα πιστοποιητικό βουλγαρικό, αλλά το Δημαρχείο της χώρας της αρνήθηκε να το κάνει για μια ακόμη φορά γιατί οι λέσβιες μητέρες δεν υπάρχουν στον βουλγαρικό νόμο. Υπήρξε αναφορά και το διοικητικό δικαστήριο είπε ότι θα πρέπει να εκδοθεί το πιστοποιητικό και να μείνει κενό ε, το σημείο στο οποίο αναφέρεται το όνομα του πατέρα. Ε, γι' αυτό και η μητέρα τώρα θα πρέπει ε, να κάνει δήλωση συγκεκριμένη για τον πατέρα. Ε, η Βουλγάρα μητέρα λοιπόν πήρε το πιστοποιητικό γέννησης, πήρε ένα νέο διαβατήριο και πήγε στη Βουλγαρία ε, χωρίς την άδεια και χωρίς ε, την γνώση της Δανέζας μητέρας. Το 18 ξεκίνησε λοιπόν μια δικαστική διαδικασία με τα αντίστοιχα δίκτυα στήριξη στη Βουλγαρία και στη Δανία έτσι ώστε να υπάρξει για την Δανέζα μητέρα πρόσβαση στο παιδί και να υπάρξει επικοινωνία αλλά το ε, Βουλγαρικό Δικαστήριο είπε ότι κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο και τα δικαιώματα των παιδιών εδώ έρχονται σε βασική αντίδραση με, την, με τους κανόνες δημόσιας τάξης της χώρας. Η τελευταία περίπτωση είναι ότι είναι τελικά επίγον να υπάρξει η αμοιβαία αναγνώριση των επισήμων εγγράφων, όχι μόνο σε επίπεδο τύπου, μορφής, αλλά και περιεχομένου, έτσι ώστε να αποφεύγονται ε, μακρόχρονες ε, διαδικασίες ε, από τις οποίες περνούν οι οικογένειες. Και στο τέλος βλέπουμε εδώ και το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών για την ιδιωτική και τη δημόσια ζωή, ε, του Οκτωβρίου υπάρχουν οι οικογένειες αυτές, ε, οι λεγόμενες οικογένειες ε, του ουρανίου τόξου, είτε αναγνωρίζονται είτε όχι. Και είναι κρίσιμο και επίγον το νομικό μας σύστημα να αναγνωρίσει την πραγματικότητα αυτή και τα κράτη-μέλη να κάνουν προσπάθεια για να θέσουν τέλος στις διακρίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Και εσείς μας κάνατε να βιώσουμε αυτές τις πάρα πολύ, πολύ πολύπλοκες καταστάσεις που δημιουργούν ανισότητες και για τα παιδιά εναντί άλλων παιδιών αλλά και ανισότητες σε σχέση με το στερικό της οικογένειας των παιδιών απέναντι στους γονείς. Σίγουρα θα υπάρξουν ερωτήσεις και αντιδράσεις. Λοιπόν, χωρίς χρονοτριβή, να δώσουμε το λόγο στην τέταρτη ομιλήτρια, την ε, δόκτωρα Αντρέα Σούλτς. Ε, είστε ε, υπάλληλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Δικαιοσύνης. Είστε αρμόδια για την αναδιατύπωση του κανονισμού Βρυξέλλες 2α και επίσης είστε και πρώτη ε, γραμματέας ε, στην διάσκεψη της Χάγκης. Είχατε περί απόσπαση. Έτσι λοιπόν είστε εμπειρογνώμενας για όλα αυτά τα θέματα και είστε και διευθύντρια της ε, κεντρικής αρχής στη Γερμανία. Σας δίνω το λόγο και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ για να μοιραστείτε μαζί μας τις γνώσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν θα ήθελα φυσικά εκ μέρους της Επιτροπής και εκ μέρους της ε, ε, την ε, Επιτροπή Τζούρι και την Επιτροπή για την Δικαιώματα του Παιδιού με τους οποίους έχουμε πολύ καλή συνεργασία και βρίσκομαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω σήμερα σε σχέση με τη διαδικασία αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλε 2α. Ένα κανονισμό που μα ενδιαφέρει πολύ και εμά, αλλά όπω γνωρίζω και εσά. Όπω βλέπετε στην πρώτη διαφάνεια, εδώ έχουμε μια γενική επισκόπηση του κανονισμού και βλέπουμε ότι πραγματικά δεν ρυθμίζει θέματα επί της ουσίας, απλώς ρυθμίζει ζητήματα δικαιοδοσίας σε, σε ό,τι αφορά ζητήματα, ε, για παράδειγμα, γαμικών ε, ε, υποθέσεων, δηλαδή διαζυγίου, χωρισμού και ούτω καθεξής, αλλά και σε ό,τι αφορά το ζήτημα που συζητάμε σήμερα εδώ, δηλαδή ζήτηματα γονικής μέρημνας όπως επιμέλειας, δικαιώματος επικοινωνίας, και ούτω καθεξής επιτροπίας ε, και ούτω καθεξής και επίσης ε, ρυθμίζει και τα ζητήματα ε, της Διεθνούς απαγωγή παιδιών με βάση την σύμβαση της Χάγης. Επίσης εδώ λάβαμε υπόψη μας για να διατυπώσουμε την πρόταση όχι μόνο τη δημόσια ακρόαση, αλλά και τις διάφορες αναφορές που έχουν αποσταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα παράπονα προς την Επιτροπή. Επίση, ήρθαμε σε επαφή με τα κρατημέλη και τις κεντρικέ αρχέ ε, και βέβαια υπάρχουν ετήσιες ε, συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα με αυτές τις κεντρικέ αρχές και διμερεί επαφέ που λαμβάνουν, που λαμβάνουν χώρα σε ό,τι αφορά δύσκολε περιπτώσει, δύσκολε υποθέσεις. Και αξιοποιήσαμε λοιπόν και αυτές τις επαφές για να διαπιστώσουμε πού τα πράγματα δεν πάνε καλά, πού δεν εφαρμόζεται, δεν εκτελείται σωστά ο κανονισμός ε, και πού μπορούν να υπάρξουν βελτιώσει. Και εδώ βλέπετε έξι τομεί του οποίου εντοπίσαμε. Ε, σε ό,τι αφορά τι ε, περιπτώσει απαγωγή παιδιών, θέλουμε να κινούνται ταχύτερα διαδικασίες και θέλουμε να υπάρχει και ένα ουσιαστικό δικαίωμα ακρόαση του παιδιού μέσα σε ένα τέτοιο, σε μια νομική πράξη τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Επίσης, η κατάργηση του εκτελεστήριου τίτλου, του ΕΞΑΚΑΤΟΥΡ. επίση η εκτελεστότητα, η εκτέλεση των ίδιων των αποφάσεων που είναι ένα ζήτημα που ρυθμίζεται στην Εθνική Νομοθεσία σήμερα. Ε, επίση, το ζήτημα τη τοποθέτηση του παιδιού σε ένα κράτο μέλο που δεν ευθυγραμμίζεται πλήρω ακόμα με την ε, πρακτική. Και επίση, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την δυνατότητα συνεργασία μεταξύ των κεντρικών αρχών διασυνοριακά. Εάν ε, λοιπόν τώρα μια ματιά στι ε, βελτιώσει αυτέ που προσπαθούμε να κάνουμε, συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τι απογέ, θέλουμε οι διαδικασίε να είναι ταχύτερε και η Επιτροπή έχει προτείνει μια διαδικαστική εναρμόνιση. Δηλαδή, τα αρμόδια δικαστήρια για τέτοιου είδου σε περίπλοκε υποθέσει θα πρέπει να είναι λιγότερα σε κάθε κράτο μέλο και επίση ο αριθμό ε, των προσφυγών θα πρέπει να είναι μικρότερο. Ε, πράγμα το οποίο δεν βρίσκει ιδιαίτερα σύμφωνα τα κράτη-μέλη. Όχι επί τη αρχή, γιατί τα περισσότερα κράτη-μέλη αποσκοπούν σε κάτι τέτοιο, αλλά για του λόγου τη επικουρικότητα. Επίση, εμεί ε, προτείνουμε διαμεσολάβηση, γιατί βέβαια φιλικοί διακανονισμοί μεταξύ των ίδιων των γονέων με τη βοήθεια διαμεσολαβητών είναι είναι λύσεις πιο βιώσιμες και ε, μακροπρόθεσμα βοηθούν και το ίδιο το παιδί. Τώρα, η ακρόαση του παιδιού είναι ο πιο φιλόδοξος στόχος μας ε, και βλέπετε για πρώτη φορά κάτι που αναφέρεται σε κόκκινο μέσα σε αυτή τη διαφάνεια. Δηλαδή, το αναφέρουμε σε κόκκινο γιατί το Συμβούλιο ήδη αποφάσισε ότι ναι, αυτό θα εγκριθεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί είπαμε ότι ναι, ισχύει ο χάρτη και των Ηνωμένων Εθνών αλλά και τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά όλα αυτά ε, τα ε, τα νομοθετήματα δεν ε, προβλέπουν ακριβώ αυτέ τι διαδικαστικέ εγγύησει στα κράτη-μέλη. Ενώ τώρα με, την, με τον νέο κανονισμό ακριβώ υπάρχει δυνατότητα αξίωση ε, του δικαιώματο από το παιδί για να γίνει ακρόαση του, ε, όπως αυτό θα προβλέπεται μέσα στην Εθνική Νομοθεσία. Άρα λοιπόν ουσιαστικά η διαφορετική μέθοδο, για παράδειγμα, που εφαρμόζεται από τα διαφορετικά δικαστήρια στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την ακρόαση του παιδιού, δεν θα μπορεί πλέον να ισχύει ω λόγο για την απόρριψη μια τέτοια ε, απόφαση. Σε ό,τι αφορά την κατάργηση τώρα του εκτελεστήριου τίτλου τη Εξεκουάρτουρ, κάτι που πρότεινε η Επιτροπή, και επ' αυτού έχουν συμφωνήσει τα κράτη-μέλη ότι ναι, θα εγκριθεί και χρειαζόμαστε και ενίσχυση των σχετικών διαδικαστικών εγγυήσεων σε ό,τι αφορά ειδικότερα την ε, υπεράσπιση. Αλλά επί της αρχής υπάρχει συμφωνία ε, και σε ό,τι αφορά ε, την ίδια την νομοθεσία δηλαδή η οποία θα εφαρμόζεται σε επίπεδο εθνική νομοθεσία σήμερα, προβλέπουμε ελάχιστη εναρμόνιση σε ό,τι αφορά του λόγου άρνηση τη εκτέλεση μια απόφαση. Γιατί τη σήμερα ημέρα δυστυχώ, όπου χρειαζόμαστε αυτή την δήλωση τη εκτελεστότητα, δηλαδή τον εκτελεστήριο τίτλο του εξεκάτου, βρισκόμαστε αντιμέτωποι συχνά ε, με ε, τι περιπτώσει εκείνε όπου ε, μία απόφαση από άλλο κράτο μέλο ε, θεωρείται ως εκτελεστή, αλλά τελικά δεν εκτελείται στην ε, πράξη, γιατί, για παράδειγμα, οι λόγοι σε ό,τι αφορά την ε, λήψη περαιτέρω μέτρων είναι λιγότεροι, για παράδειγμα, στο δεύτερο κράτος μέλος, σε ό,τι αφορά δηλαδή συγκεκριμένα προστατευτικά μέτρα. Άρα, λοιπόν, εδώ κάνουμε μια ελάχιστη εναρμόνιση, με βάση την οποία τα κράτη-μέλη μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν την εθνική του ομοθεσία, εφόσον παραμένει συμβατή με τον κανονισμό. Ε, τώρα, σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του παιδιού, έχουμε δύο νέα μέτρα. Ε, καταρχήν έχουμε τα εκπαιδευτικά μέτρα, γιατί βέβαια αυτοί οι κανόνες έχουν προβλεφθεί για την περίπτωση όπου ε, χρειάζεται ε, νέους γονείς ε, το παιδί και η υιοθεσία για παράδειγμα δεν είναι το κατάλληλο εργαλείο για κάτι τέτοιο. Διαπιστώσαμε όμως ότι υπάρχει ότι ένα διαφορετικό ένας διαφορετικός τύπος τοποθέτησης αφορά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Δηλαδή ε, εκπαιδευτικού χαρακτήρα τοποθέτηση. Ένα παιδί δηλαδή το οποίο ε, επιδεικνύει μια ε, παραβατική συμπεριφορά και μπαίνει ακριβώς σε μια τέτοια διαδικασία εκπαιδευτικών μέτρων έτσι ώστε να επανέλθει εντό εισαγωγικών. Αυτό λοιπόν είναι τελείως διαφορετικό από την τοποθέτηση ενός παιδιού σε μια νέα οικογένεια. Επίσης υπάρχει και μια περίπτωση όπου για παράδειγμα ένα παιδί διαβεί σε, μια, σε ένα κράτος μέλος ε, και θα πρέπει να βρεθεί μια νέα οικογένεια για αυτό το παιδί, αλλά συγγενείς αυτού του παιδιού θα βιούν σε άλλο κράτος μέλος. Και για αυτή λοιπόν την περίπτωση προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Ε, και για να υπάρξει βέβαια εκτέλεση όλων αυτών χρειαζόμαστε και συνεργασία μεταξύ των ε, κεντρικών αρχών. Υπάρχουν δηλαδή ε, ζητήματα ε, που είχαν προκύψει σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ε, αλλά με τον γενικότερο κανονισμό για την προστασία των δεδομένων που εγκρίθηκε είναι ακόμα σημαντικότερο να υπάρχουν σαφείς κανόνες και να εφαρμόζονται σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων. Και καθώ βέβαια το δικό μα πάνελ εστιάζει ειδικότερα και στο δικαίωμα επικοινωνία του γονέα με το παιδί, να σας πω ότι υπάρχει και ένα νέο θέμα που συζητείται αυτή την περίοδο ως προς την περίπτωση ε, της ε, απαγωγής ενός παιδιού. Δηλαδή όταν η διαδικασία ακόμα εκκρεμία, όταν ακόμα τρέχει το δικαστήριο δεν έχει μία δικαιοδοσία σε ό,τι αφορά την ίδια την επιστροφή, αυτό το δικαστήριο ενθαρρύνεται να εξετάσει κατά πόσο ε, θα πρέπει να ισχύσει ένα δικαίωμα επικοινωνίας ενώ το συνεχίζεται η απαγωγή του παιδιού, έτσι ώστε να μην χαθεί επικοινωνία με τον άλλο γονέα που έχασε το παιδί. Ε, και τώρα να περάσω στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι της παρουσίασής μου, δηλαδή τα ε, επόμενα βήματα. Εργαζόμαστε λοιπόν πυρετοδός σε αυτή την περίοδο και ε, ελπίζουμε πως την επόμενη εβδομάδα θα είναι η τελευταία συνάντηση σε επίπεδο κορεπέρ στον τομέα ΔΕΗ, έτσι ώστε η Αυστριακή Προεδρία να παρουσιάσει αυτή την πρόταση στις 7 ε, Δεκεμβρίου, ε, ώστε το Συμβούλιο να καταλήξει σε ένα γενικό προσανατολισμό σε ό,τι αφορά τα σχετικά άρθρα με τις σχετικές ε, αιτιολογικές σκέψεις. Και από εκεί και μετά βέβαια εκκρεμούν και η οριστικοποίηση των ε, παρατημάτων, άλλων αιτιολογικών σκέψεων και ό,τι καθεξής, αλλά θα, αυτό θα το αναλάβει η Ρουμανική και, ε, Προεδρία και η νωρίτερη προθεσμία που προβλέπουμε ε, για την εφαρμογή, την ειδική εφαρμογή αυτού του κανονισμού είναι η 1η Ιουλίου του 2022. Αλλά αν κοιτάξω τα τρία χρόνια που περάσαν και τα οποία εξετάζαμε αυτό το κανονισμό, περάσα πολύ γρήγορα και νομίζω και ο υπόλοιπο καιρό θα περάσει και αυτό πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε για την βούλησή σα ε, να επιταχύνετε τις διαδικασίες, ε, να τις αποσαφηνίσετε και να προωθήσετε τη διαμεσολάβηση. Ελπίζω ότι εκ περιτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, ε, οι Προεδρίες μάλλον, ε, δεν θα καθυστερήσουν, ούτε θα ανακόψουν τον, την αποφασιστικότητά σας. Μου δίνετε πολύ μεγάλες ελπίδες. Σας ευχαριστώ πολύ για όλο αυτό το έργο. Λοιπόν, ανοίγω τώρα τη συζήτηση. Έχουμε 10 λεπτά, Πρόεδρε, για τις ερωταπαντήσεις. Ποιος ε, θα ήθελε να πάρει το λόγο. Δυστυχώς μόνο 10 λεπτά έχουμε στην ε, διάθεσή μας, γιατί ακόμα έχουμε δύο πάνελ και θα μπορέσετε να ξαναπάρετε το λόγο. Ποιος θέλει τώρα το λόγο, παρακαλώ. Αν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ε, και εγώ είμαι δικηγόρος ε, στις, στο δικηγορικό σύλλογο των Βρυξελών. Θα ήθελα να αναφερθώ ε, σε παιδιά που προέρχονται από τις άκρως αποκεντρωμένες περιοχές και στο Βρυξέλλες 2α δεν λαμβάνεται υπόψη η απόσταση και ως ε, δικηγόρος ε, δεν μπορούμε να καταλάβει κάποιος ότι ε, φεύγει κάποιος τη Δευτέρα, φτάνει την Τρίτη και φτάνει, το χάρη, ε, στη Γαλλία. Έτσι λοιπόν θέλω να απευθυνθώ στην Κομισιόν. Έχουμε παιδιά που είναι σε δυσκολία, που βρίσκονται ουσιαστικά με απαιτήσει επιστροφής και είναι σε μια αδύνατη κατάσταση και τα δικαστήρια δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη διευκρίνησή σας. Είναι πολύ σημαντικό και στην Γουιάννα και με τις ε, χώρες ε, που είναι γύρω ε, από αυτό το διαμέρισμα ότι γίνεται από πολύ πολύπλοκη κατάσταση. Σας ευχαριστώ λοιπόν που επισημάνατε αυτό το θέμα. Υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Δεν βλέπω. Ευχαριστούμε λοιπόν, Μπέτ. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Μήπως θα μπορούσαμε να ζητήσουμε μία απάντηση από την κυρία Σούλτς για τις άκρως αποκεντρωμένες περιοχές, Πρόεδρε. Διαβάσαμε στα μάτια σας ότι κατανοείτε πολύ καλά την κατάσταση. Αλλά μήπω μπορείτε και να μας το εκφράσετε, μην διστάζετε παρακαλώ να σηκώσετε και το χέρι και να ζητήσετε το λόγο. Κοιτάξτε, δεν είμαι γνωστή <laughs> για την ντροπαλοσύνη μου. Γνωρίζουμε το πρόβλημα όμως. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό το πρόβλημα προκαλείται από το ουσιαστικό και γενικό δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου γιατί οι κανόνες περί δικαιοδοσίας κρίνουν μόνο σε ποιο κράτος μέλος πρέπει να δικαστεί μία υπόθεση και αν είναι η Γαλλία δεν θα αποφασίσει το ενωσιακό δίκαιο που στη Γαλλία και ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο της απόφασης. Ξέρω βέβαια ότι οι συνάδελφοι μας από τον Οργανισμό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Συμβουλίο της Ευρώπης εργάζονται προκειμένου να δημιουργήσουν μια ευαισθητοποίηση για το θέμα αυτό και να τροποποιήσουν και το ουσιαστικό δίκαιο προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν σε, όπως και σε άλλα θέματα. Ε, που αφορούν το νοσιακό δικαίωμα δεν θα ήταν δυνατό να βάλουμε το θέμα της απόστασης γιατί αν ε, κατοικεί κάποιος στην Καλυδονία χρειάζεται 22 ώρες να επιστρέψει στην Γαλλία ενώ στην Πολυνησία 24 ώρες. Ίσως ε, λοιπόν και η απόσταση θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη στα δικαστικά πρακτικά. Δεν ζητεί άλλο το λόγο. Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε λοιπόν στο δεύτερο πάνελ. Πάνω κάτω έχουμε σεβαστεί και το χρόνο. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές που ήταν πολύ ακριβείς και ήταν και πολύ ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσεις. Τώρα θα παρουσιάσουμε τις βέλτιστες πρακτικές ε, σε ό,τι αφορά ε, την ακρόαση του παιδιού επέμενε ήδη στο θέμα αυτό, το πρώτο πάνελ, δηλαδή να δούμε ποιες είναι οι πρακτικές ε, στις ε, διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες ε, σε σχέση με τις διασυνοριακές γονικές διαφορές και την ακρόση του παιδιού. Και φυσικά τα δικαιώματα του παιδιού προστατεύονται σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες. Έχουμε και τις Εθνώση σε σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού. Βέβαια, ε, θέλουμε να δούμε τι γίνεται και στην πράξη. Έχουμε τρεις συμπειρογνώμονες και θα ξεκινήσω με την ε, κυρία Θάλια Κρούγκερ, η οποία είναι καθηγήτρια σε θέμα, ε, στα θέματα ε, ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Από το 2010 είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας και συμμετέχει σε πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα στον τομέα αυτό, κυρίως σε ό,τι αφορά στην ακρόαση των ε, παιδιών που θα μας παρουσιάσετε τώρα. Και φυσικά μας ε, ενδιαφέρει πάρα πολύ να βελτιώσουμε το θέμα της ακρόασης των παιδιών. Σας ακούμε. Um, thank you very Thank you very much for Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και για την πρόσκληση. Καταρχήν θα πω ότι εδώ θα παρουσιάσω κάποια προκαταρκά αποτελέσματα του προγράμματος Voice. Είναι ένα πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι εταίροι μας είναι το Missing Children Europe, το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας της Γένοβας και της και το κέντρο ΙΚΟ. Πολλοί από τους εταίρους μας βρίσκονται στην αίθουσα επίσης σήμερα και τους ευχαριστώ για τη συνεργασία. Και θέλω να ευχαριστήσω και τους ερευνητές των Πανεπιστημίων της Αμβέρσας και της Γένοβας για το νομικό τους έργο, για αυτό το πρόγραμμα. για να ξεκινήσω με το τι κάναμε. Αναλύσαμε την ομολογία από την 1η Μαρτίου 2005 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017. Η 1η Μαρτίου είναι ημερομηνία θέσεων σε ισχύ κανονισμού Βρυξέλλες 2α, γι' αυτό έχουμε αυτή την ημερομηνία και τελευταία ημερομηνία. Ουσιαστικά αφορά την ημερομηνία, οπότε ξεκίνησε το ερευνητικό μας έργο. Εξετάσαμε 938 υποθέσεις ε, από αυτά τα κράτη-μέλη. Δεν μπορέσαμε να συμπεριλάβουμε όλα τα κράτη-μέλη λόγω χρηματοδότησης. 8 αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και 54 υποθέσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και είδαμε τις αποφάσεις ε, και πώς σχετίζονται με το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, πώς επίσης το βέλτιστο συμφέρον συνδεόταν εκ νέου με άλλα νομικά μέσα. Έτσι λοιπόν το πρόγραμμα ήταν πιο ευρύ από το θέμα της ακρόασης του παιδιού, λαμβάνει υπόψη το συμφέρον του παιδιού και ως μέρος αυτού την ακρόαση του παιδιού. Εργαστήκαμε με τους δικούς μας ερευνητές και τους εθνικούς αντιποκριτές για τις γλώσσες που δεν καταλαβαίναμε και τι είδαμε, ότι τα δικαστήρια με, ε, χρησιμοποιούν με διάφορο τρόπο την έννοια βάλτιση στο συμφέρον του παιδιού. Μερικές φορές ε, Απλά λένε ότι οι συμβάσει δεν κοιόνται τα συμφέροντα του παιδιού και το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Δεν χρειάζεται λοιπόν ε, πολύ συγκεκριμένα να το διερευνήσουμε αυτό για ένα συγκεκριμένο παιδί και σε κάποιε περιπτώσει συνδέονταν το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού με ε, τι Βρυξέλλε 2 και την σύμβαση τη Χάγη ε, για του λόγου που υπάρχουν εκεί, στο βαθμό δηλαδή που λέγεται ότι η σύμβαση εγγυάται τα δικαιώματα έτσι. Και είχαμε κάποιες περιπτώσεις όπου το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού συνδεόταν με τους λόγους για την εξαίρεση, δηλαδή το κίνδυνο να, να, μάλλον, να, να τεθεί το παιδί σε κίνδυνο ή να βρεθεί σε μια παράδεκτη κατάσταση. Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού στις περισσότερες περιπτώσεις έκανε τις εξαιρέσεις ευρύτερες και κάποιες, ε, σε κάποιες υποθέσεις ε, θεωρήθηκε το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού μια ανεξάρτητη έννοια δίπλα από αυτά τα νομικά μέσα. Έτσι λοιπόν οι αναφορές ε, στο βελτίστο συμφέρον του παιδιού όταν γίνονταν ρητά λάμβαναν ε, εδώ έχουμε, έχουμε κάνει έρευνα και στις, ε, στις αναφορές που υπονοούνται όμως υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος που συνδέεται η ρητή αναφορά στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού με συγκεκριμένο έγγραφο. Στις περισσότερε περιπτώσεις συνδέεται με το άρθρο 3.1 της Σύμβασης του ΙΕ σε 367 περιπτώσεις με τη Σύμβαση για την Απαγωγή των Παιδιών, σε 32 περιπτώσεις, σε άλλα διεθνή νομοθετήματα. Ε, είχαμε διάφορες πράξεις ε, που αφορούν το οικογενειακό δίκαιο ή την εθνική νομοθεσία. Σε 26 περιπτώσεις αναφέρθηκα συγκεκριμένα στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι 16 από αυτές 26 υποθέσει ε, ε, αναφέρθηκαν στην ε, απόφαση από το Λετωνικό Δικαστήριο. Νομίζω ότι είναι καλό που αναφέρθηκε σε αυτό το δικαστήριο. Και τι είδαμε, ότι σε ορισμένε περιπτώσει κάποια εθνικά δικαστήρια εξακολουθούσαν να παραβαίνουν στην ε, υπόθεση Νόιλι. Αν ε, δείτε και τους εμπειρογνώμενους που εργάζονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αυτοί θα πούνε ότι είχαμε ουσιαστικά την υπόθεση της Λετωνίας ε, που έρχονταν σε αντίθεση με τον Όλιγκερ. Και πάλι βλέπουμε ότι οι εθνικές υποθέσει παραπέμπουν περισσότερο στην υπόθεση Νόλιγκερ παρά στην υπόθεση της Λετωνίας. Και 32 υποθέσεις αναφέρονται σε άλλη νομολογία, γιατί αναφέρθηκαν και σε αλλοδαπή νομολογία, παραδείγματο χάρη σε πολλέ ε, υποθέσει του Ηνωμένο Βασίλειο. Τρει αναφέρθηκαν στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεν περίεργο γιατί δεν έχουμε πολλέ υποθέσει εκεί. Και ε, Έχουμε και άλλους λόγους αναφορά στο βελτιστά συμφέρον του παιδιού, όπως είναι η νομική βιβλιογραφία. Τι βλέπουμε στις αναφορές ε, που έγιναν. Κάποια δικαστήρια είπαν ε, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και η ανάλυση θα πρέπει να αφορά τη χώρα της συνήθως κατοικίας. Στην πραγματικότητα, θα πρέπει να είναι ε, εντός της ευρωπαϊκής διαδικασίας, όμως κάποια δικαστήρια δεν το κάνουν. Ε, λένε ότι αυτό πρέπει να το κρίνει το δικαστήριο της σύντουσης κατοικία. Επίσης, το δικαστήριο λέει ότι βέλτιση των συμφέρον σημαίνει μια ταχύ επιστροφή. Δεν το λένε πάντα αυτό. Γιατί κάποια δικαστηρία λένε όχι, αλλά χρειαζόμαστε κάποιο χρόνο για να προετοιμαστεί η επιστροφή του παιδιού. Ε, εδώ βλέπουμε δικαστήρια που ε, λαμβάνουν υπόψη το θέμα της ενίσχυσης του μεμονωμένου παιδιού και το δικαστήριο λέει σωστά νομίζω ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού είναι πιο σημαντικό από το να τιμωρηθεί ο γονέας ε, για το λάθος που έκανε και το βέλτιστο συμφέρον ε, θα πρέπει να συνδέεται με το μεμονωμένο παιδί και να μην έχουμε μια γενική έννοια, αλλά να κοιτάμε την υπόθεση ενός συγκεκριμένου παιδιού. Μερικές φορές συνδέεται με το κράτος της συνήθους κατοικίας, ε, μερικές φορές μπορεί να συνδέεται με το θέμα ε, του καταφυγίου. Επίσης μπορούμε να δούμε αν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, ε, δηλαδή να βρεθεί το παιδί σε μια παράδεκτη κατάσταση ή να αντιμετωπίσει το παιδί βία, είτε ψυχολογική είτε σωματική. Τα δικαστήρια επίσης λένε ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού είναι το να λάβουμε υπόψη την ε, άποψη του παιδιού, τη γνώμη του παιδιού και έχουμε το θέμα της ακρόασης. Δηλαδή να δούμε τι ακριβώς λέει το παιδί για τα δικά του, για το δικό του βέλτιστο συμφέρον. Επίσης ε, υπάρχει και το θέμα της ε, διαφοράς μεταξύ των γονέων. Ε, και λένε πολύ σωστά στο δικαστήριο ότι μπορεί να προκαλούνται περισσότερα προβλήματα ε, γιατί αυτή η σύγκρουση μεταξύ των γονέων δεν είναι κάτι καλό για το παιδί. Επίσης, ε, το καλύτερο συμφέρον του παιδιού είναι μια κατηγορία γραμμή σε όλες τις περιπτώσεις και κατόπιν ζυγίζονται τα δικαιώματα του παιδιού και των γονέων. Όλα αυτά τα ζητήματα, λοιπόν, τα βλέπουμε στην ομολογία. Εδώ βλέπετε μία σειρά ε, παραγόντων που προωθούν ε, αριστερά τα των συμφέρον ε, και στην άλλη στήλη έχουμε τους αρνητικούς παράγοντες. Όλα αυτά τα έχουμε πάρει από την ομολογία. Θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρον ότι ο κατάλογος των αρνητικών παραγόντων είναι πιο μακροσκελής από ότι ο κατάλογος των θετικών. Δηλαδή, φαίνεται είναι εύκολο να πούμε ότι η κακομεταχείριση δεν είναι προ το βαλτιστό συμφέρον του παιδιού, όμω ε, το θέμα είναι ότι είναι δύσκολο να βρούμε τι είναι προ το βαλτιστό συμφέρον του παιδιού. Έτσι λοιπόν, τα δικαστήρια τι λένε, ε, είναι ότι εξετάζουμε την ευημερία του παιδιού, όμως τι σημαίνει αυτός ο όρος ευημερίας, εμείς δεν ξέρουμε ως δικηγόροι. Όμως, ε, από την άλλη πλευρά έχουμε και την έρευνα των κοινωνιολόγων, και κατόπιν ε, συσχετίζουμε αυτά τα δύο για να δούμε αν δικηγόροι κατανοούν ορθά τον όρο ευημερία. Ε, είναι διατήρηση ε, των σχέσεων στην οικογένεια, το να επιστρέψει μαζί με τον γονέα που έκανε την απαγωγή, αν υπάρχει ένας ισχυρός δεσμό. δηλαδή ο νέο μπορεί να πάει μαζί με το παιδί. Αυτό θεωρείται θετικό για το βέλτιστο συμφέρον και επίση εξετάζουν τα δικαστήρια την ε, ανάπτυξη του παιδιού σε ένα ασφαλές περιβάλλον, την ψυχολογική του, ψυχοκοινωνική του ανάπτυξη και αν υπάρχουν ικανοποιητικές ε, συνθήκες διαβίωσης. Όταν λέει ικανοποιητικές, το δικαστήριο ξεκαθαρίζει ότι δεν θεωρεί ότι απλώς πρέπει να είναι λίγο καλύτερες ή χειρότερες συνθήκες από ό,τι στην άλλη χώρα. Αν δείτε τους αρνητικούς παράγοντες, κάτω-κάτω βλέπετε ε, ότι η έλλειψη εργασίας ή ε, τα προβληματική οικονομική κατάσταση δεν είναι προς το βαλτιστό συμφέρον του παιδιού, αλλά θα πρέπει να ζυγίσει κανείς που είναι καλύτερες συνθήκες. Πάμε στην επόμενη, αφορά, στην επόμενη διαφάνεια που αφορά την ακρόαση. Εμείς βρήκαμε 194 υποθέσεις όπου υπήρχε συζήτηση για το θέμα της ακρόασης του παιδιού για το πώς αυτό μπορεί να συνεισφέρει στο βελτιστό συμφέρον του παιδιού. Των 26 υποθέσεις ε, το παιδί δεν ακούστηκε και υπήρξε μια εξήγηση γιατί. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε πολλές υποθέσεις, ότι δεν ξέρουμε αν ε, υπήρξε ακρόαση ή όχι του παιδιού, δεν ξέρουμε τι έκανε το δικαστήριο, ούτε καν τι είπε το παιδί. Στην έρευνά μα δεν μπορούμε να το δούμε αυτό, γιατί εμείς εξετάσαμε την ομολογία. Για αυτές τις 194 υποθέσεις είδαμε ότι ενίοτε η ακρόαση είχε στόχο ε, να δει αν το παιδί είναι ενάντια στην επιστροφή. Όμως, πολλές φορές η ακρόαση πήγε πιο μακριά. το χάρη, να ακούσουμε το παιδί για να δούμε αν υπάρχει κίνδυνος υπάρχει κίνδυνος για το παιδί για να επιστρέψει. Ας ακούσουμε το παιδί και να το δούμε από την οπτική του παιδιού. Ακόμη και αν ε, αυτό μπορεί να μην σημαίνει απαραίτητα ότι ε, αντίκειται το παιδί στην επιστροφή και αυτό είναι συγκεκριμένο λόγο άρνηση. Επίση, να δούμε αν έχει εγκατασταθεί το παιδί στον περιβάλλον, να έχει εγκληματιστεί. Και πολλές ε, φορές είχαμε και αντίρρηση αλλά και κίνδυνο για το παιδί που συνδυαζόταν όταν δεν είχαμε ακρόαση του παιδιού. Θεώρησα ενδιαφέρον ότι πολλά δικαστήρια εξήγησαν γιατί δεν άκουσαν το παιδί και εγώ νομίζω ότι αυτό οφείλει στον κανονισμο βρυξελλης Βρυξέλλες 2α και στη δουλειά της Κομισιόν πραγματικά μου τονίσει το θέμα της ακρόασης του παιδιού. Αν ε, τα δικαστήρια δεν ακούνε το παιδί θα πρέπει τουλάχιστον να εξηγήσουν γιατί όχι. Ο κύριος λόγος ε, προφανώς ε, είναι η ηλικία. Ξέρουμε ότι πολλές φορές ε, τα παιδιά που απάγονται είναι πολύ μικρά, μπορεί να είναι κάτω των δύο ετών. Όμως μπορεί μερικές φορές τα παιδιά να εκφράσουν και την άποψή τους με άλλους τρόπους, όχι με λόγια. Έτσι λοιπόν θα έλεγα ότι είναι σκόπιμο να ακουστεί το παιδί κυρίως σε περιπτώσεις όπου το παιδί δεν μπορεί να εκφραστεί καλά επειδή μπορεί να υπάρχει ένα πρόβλημα ή να έχει μια ασθένεια. Ε, σε άλλες περιπτώσεις ε, κάποιο άλλο όργανο μπορεί να άκουσε το παιδί. Είπε το δικαστήριο θα πρέπει να ακούσει το παιδί το άλλο δικαστήριο στην άλλη χώρα. Όμως ε, βέβαια το τι είπε στο πρωτοδικείο το παιδί δεν σημαίνει ότι επανέλαβε τα ίδια και στο επόμενο δικαστήριο. Επίσης, ε, μπορεί να υπάρχει ένα ε, τραύμα και δεν κρίνεται σκόπιμο να ακούσουν το παιδί. Θεωρείτε λοιπόν ότι δεν είναι απαραίτητο στην περίπτωση αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Μας ε, δείχνετε πώς το θέμα της ακρόσεως του παιδιού είναι κάτι πολύ χρήσιμο στις περισσότερες περιπτώσεις και πρέπει να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει αυτό στα πολύ μικρά παιδιά, στα πολύ νεαρά παιδιά. Και το ότι αιτιολογείται ε, ακόμη και εκτελεούνται για περιπτώσει όπου δεν υπάρχει ακρόαση του παιδιού και αυτό πηγαίνει προς ε, τις, ε, τη δική μας πρόθεση. Στη συνέχεια θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Φρασίσκο Χαφιέ Φορκάντα Μιράντα. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Είστε ε, αρμόδιος επικεφαλής στο ε, Διεθνές Δίκτυο Δικαστών. Επίσης, έχετε εργαστεί στο εφετείο της Μαδρίτης και είστε εκπρόσωποι της Ισπανίας στο Διεθνές ε, Δίκτυο Δικαστών στη Χάγη έχει και το σημείο επαφής ε, για εμπορικές και αστικές υποθέσεις ε, για την ε, Ισπανία. Και εσείς έχετε περίπου 15 λεπτά στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Δεν μπορώ μέσα σε 8 λεπτά να κάνω την παρουσίασή μου. Ζητώ συγγνώμη και από τους διευμηνείς δεν έχω τον απαιτούμενο χρόνο. 15 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας, όχι 8 λεπτά. Οπότε μπορείτε να κάνετε την παρουσίασή σας και μετά θα περάσουμε στις ερωταπαντήσεις, όπως και με τους προηγούμενους συναδέλφους σας. Θα προσπαθήσω να εκθέσω κάποιες ιδέες τις οποίες θεωρώ σημαντικές. Πριν ξεκινήσω με την παρουσίαση, θα ήθελα να αναφερθώ στην ιδέα την οποία εγώ θεωρώ ουσιώδη. Έχω το ειδικό χαρακτηριστικό να είμαι δικαστής σε επίπεδο οικογενειακών διαφορών στη χώρα μου για αρκετά χρόνια και ασχολήθηκα με πάρα πολλά παιδιά και αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει κανείς να εξετάσει, ε, να, να ακούσει έναν ανήλικο ιδιαίτερα κάτω από δραματικές συνθήκες και ιδιαίτερα όταν έχουν ξεκινήσει ήδη δικαστικές διαδικασίες. Σε διεθνές επίπεδο υπάρχουν κάποια διεθνή στάνταρ για την ακρόαση των παιδιών, ιδιαίτερα στο άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα παιδιά, για τα δικαιώματα των παιδιών. Και έχουμε επίσης και το άρθρο 24 της Χάρτας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά αυτοί οι κανόνες είναι δύσκολο να μεταφερθούν στην πραγματικότητα. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών λέει ότι το παιδί θα πρέπει να μπορέσει να εκφραστεί και κάτω από ποιες συνθήκες, αλλά στην πραγματικότητα εμείς φαίνεται ότι δεν επιτυγχάνουμε να οργανώνουμε με σωστό τρόπο τις ακροάσεις των ανηλίκων. Στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης είχα την δυνατότητα να εκπροσωπήσω τη χώρα μου για αρκετά χρόνια στην Επιτροπή Δικαστικής Συνεργασίας, Νομικής συνεργασία όπου συζητήσαμε το θέμα των λεγόμενων κατευθυντηρίων γραμμών ε, child friendly, φιλικών για τα παιδιά. Και είχαμε συζητήσει το πώς θα αντιμετωπίζουμε τα παιδιά όταν έχουν ε, επαφή με την δικαιοσύνη. Και τελικά η πραγματικότητα στις διάφορες χώρες οι οποίες αυτές αποφασίζουν για την επαφή αυτή, για την επικοινωνία αυτή, δείχνει η πραγματικότητα ότι σε επίπεδο θεωρητικό έχουμε κάτι το οποίο πολύ καλό είναι, αλλά σε επίπεδο πρακτικό όχι. Και νομίζω ότι είναι απαραίτητο οι διάφορες χώρες να έχουν μια ειδική νομοθετική ρύθμιση για, την, για τα παιδιά και τις οικογένειες, αλλά θα πρέπει και οι εργαζόμενοι στα πλαίσια αυτών των δικαιοδοσιών, οι δικαστές λοιπά να έχουν ειδικέ γνώσεις σχετικά με τους ανηλίκους. Ο ανήλικος θα πρέπει να είναι πάντα στο κέντρο της προσοχής και τα συμφέροντά του θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Υπάρχουν όμως κάποια εμπόδια σε πολιτισμικά θα έλεγα και σε επίπεδο νοοτροπίας σε σχέση με τους ανήλικους θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τους κανόνες που εμποδίζουν τη σωστή ακρόαση. Ε, αναφέρομαι επίσης και στο άρθρο 7.3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των ανθρώπων με ε, αναπηρίες. Και λέγεται ότι τα παιδιά με αναπηρίες θα πρέπει να έχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ακούσουμε τα παιδιά προσαρμοζόμενοι κάθε φορά στην αναπηρία αυτή. Απαιτείται ευελιξία και εξειδίκευση και θα πρέπει διάφορες χώρες να εφορμόζουν σωστά τις διεθνείς συμβάσεις γιατί αλλιώς αποτυγχάνουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία έχουν μεγάλη σημασία ε, ποια είναι η στιγμή οριμότητας στην οποία μπορεί να φτάσει ένας ανήλικος έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η γνώμη του. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε επί μακρόν. Αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα να πω εδώ στο Κοινοβούλιο, η ιδέα που θα ήθελα να παρουσιάσω είναι ότι δεν υπάρχουν βέβαια κάποιες απόλυτες αρχές. Ε, και ότι ακόμα και ένας ανώριμος ε, ανήλικος μπορεί να εκφραστεί με τρόπο ανώριμο, αλλά παρόλα αυτά από αυτό μπορούμε να πάρουμε στοιχεία έτσι ώστε να καταλήξουμε σε κάποιες περάσματα. Πάρα πολλές χώρες λέγουν μέσω των νομοθετικών ρυθμίσεών τους ότι από την ηλικία αυτή ο ανήλικος είναι όριμος και γι' αυτό η άποψή του θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Όμως για να ορίσουμε το πώς είναι όριμος ένας ανήλικος απαιτούνται έρευνες από πάρα πολλούς εξειδικευμένους ιατρούς, ψυχολόγους και μπορεί και 17 διαφορετικές επαγγελματικές κατηγορίες να παρέμβουν για να μπορέσουν να ορίσουν την οριμότητα ενός ανηλίκου. Οπότε αναρωτιέται κανείς, χρειάζεται να παρεμβαίνουν όλοι αυτοί έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την ακρόαση ενός ε, νέου, ενός μικρού παιδιού. Ε, στις χώρες όπου η φωνή του παιδιού ακούγεται, σε τρεις μέρες παρεμβαίνει ο ψυχολόγος, ή κοινωνικές υπηρεσίες, και εκφράζεται η άποψη. Σε άλλες χώρες η διαδικασία αυτή κρατάει έξι μήνες, από τρεις μέρες σε έξι μήνες. <clears throat> υπάρχει ε, αντιπαράθεση, υπάρχει πρώτη ακρόαση, δεύτερη ακρόαση, λοιπόν, ε, και μπλέκεται μια πολύ, ένας πολύ μεγάλος αριθμός ε, ενδιαμέσων και αυτό δημιουργεί μια διαδικασία στάθειας και ανασφάλειας. Θα πρέπει να πούμε επίσης ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ίσως δεν περιλαμβάνει οδηγίες για τη σωστή εφαρμογή των ρυθμίσεων τις οποίες προωθεί. Τώρα βρισκόμαστε στη διαδικασία μεταρρύθμισης των Βρυξελών 2α με το οποίο ασχολείται το Κοινοβούλιο. Και γι' αυτό θα ήθελα να πω ότι αν η αναθεώρηση του κανονισμού αυτού, σε αυτό το πλαίσιο, οδηγεί στο να επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά αυτά τα οποία λέει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών ή η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τόσο σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να είναι κάτι το θετικό, αλλά πραγματικά θα υπάρξει ουσιαστική βελτίωση ε, για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται ε, σε μια οικογενειακή διαφορά ένας ανήλικος πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο, ο κανονισμός να μην αλλοιώσει φυσικά την νομοθεσία που ισχύει σε κάθε χώρα, αλλά να βελτιώσουν τις ακροάσεις των ανηλίκων όταν αυτές συμβαίνουν. Το ερώτημα λοιπόν είναι το τελικό κείμενο στο οποίο θα καταλήξουμε και το οποίο σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα τεθεί σε ισχύ το 2022 θα αποτελεί μια ουσιαστική βελτίωση της ισχύουσας κατάστασης. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο τίθεται. Έχουμε τις πρακτικές οι οποίες λέγουν στον επαγγελματία το τι πρέπει να κάνει για να οργανωθεί μια σωστή ακρόαση ξεκίνησε θα έλεγα να ακούγεται ότι δεν έχουμε πρακτικούς τρόπους για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την οριμότητα μιας μαρτυρίας ενός ανήλικου. Έχουμε όμως μια λύση την οποία προτείνει το Συμβούλιο της Ευρώπης όχι ειδικά για την ακρόαση του ανηλίκου αλλά κάποιες γενικότερες συστάσεις για την αντιμετώπιση του ανήλικου όταν έρχεται σε επαφή με νοικαστικές διαδικασίες. Είναι λοιπόν σημαντικό, πιο σημαντικό από οτιδήποτε άλλο να λάβουμε υπόψη μας ότι η νομική εφαρμογή ε, των ρυθμίσεων ε, από μία χώρα έχει πολύ μεγάλη σημασία μόνο στο βαθμό κατά τον οποίο εφαρμόζεται με σωστό τρόπο προφανώς. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις στο έγγραφο το οποίο είχα ετοιμάσει. Τίθεται σαν παράδειγμα το θέμα της αξιολόγησης των μαρτυριών των ανηλίκων και υπάρχει επίσης και ειδικές, οι ξε, ξεχωριστές ιδέες για τις απαγωγές σε διεθνές επίπεδο, τις οικογενειακές. Όταν ο ανήλικος, σαν παράδειγμα, αρνείται να επιστρέψει ε, σε ποιο βαθμό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η μαρτυρία του. Αν δεν θεωρείται όριμος, η αξία την οποία έχει η μαρτυρία προφανώς μικρύνεται. Και γι' αυτό εφόσον μιλάμε για το άρθρο 13.2, ε, Αναφερόμαστε σε περιπτώσεις στα πλαίσια των οποίων ε, αναζητείται να βρεθεί πιθανότητα βίαιης κατά κάποιο τρόπο παρακράτησης ή παρεμπόδισης ε, του παιδιού να επιστρέψει στη χώρα προέλευσής τους. Υπάρχουν ε, πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες εδώ, οι οποίες μερικές φορές καθιστούν την μαρτυρία του ανηλίκου πολύ λιγότερο σημαντική. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε ότι όταν υπάρχουν τέτοιου είδους συνέπειες, όταν υπάρχουν προβλήματα οικογενειακής βίας, ε, σεξουαλικών καταχρήσεων, ε, στις περιπτώσεις απαγωγών και σε σχέση με την άποψη του ανήλικου δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, θα πρέπει όμως να ακουστεί ενώ αντίθετα όταν ένας όριμος ε, ανήλικος ε, αντιτίθεται σε μία επιστροφή, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λυθεί υπόψη. Σχετικά με την επόμενη διαφάνεια τώρα. Το δικαίωμα το οποίο έχουν τα παιδιά πρέπει να θεωρείται δικαίωμα, αλλά όταν ασκείται το δικαίωμα αυτό, έχουμε ένα πρόβλημα στα πολωνικά λέει ο η Πρόεδρος. Μπορείτε να συνεχίσετε. Θα ήθελα να πω ότι όταν ασχολούμαστε με το θέμα της ακρόασης των ανηλίκων στις εθνικές δικαστικές ε, διαδικασίες, ε, πολύ συχνά σε ορισμένες διαδικασίες, σε ορισμένες χώρες θεωρείται ότι οι δηλώσεις ε, του ανήλικου θεω... αποτελούν μία απόδειξη και μπορεί να χρησιμοθεί η απόδειξη αυτή σε μία δικαστική διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει και δυνατότητα αντιπαράθεσης και οι αντίθετοι δηλαδή θα πρέπει να μπορέσουν να ακουστούν και να αποδείξουν ότι μπορεί να απορρίψουν τον ισχυρισμό. Αλλιώς, εφόσον δεν έχουν την δυνατότητα αυτή, τότε δεν πρέπει να θεωρηθεί απόδειξη η μαρτυρία. Το θέμα είναι λοιπόν με ποιο τρόπο θα ρυθμίσουμε σε εθνικό επίπεδο την ακρόαση ενός ανηλίκου στα πλαίσια μιας δικαστικής διαδικασίας, έτσι ώστε να έχει το βάρος που απαιτείται και να μπορέσει να είναι χρήσιμη. Εδώ βλέπουμε ε, το τι συμβαίνει με την φωνή του παιδιού, ενός παιδιού στα πλαίσια των Βρυξελών 2α. Εδώ οργανώνεται η ακρόαση του ανηλίκου στα πλαίσια των διεθνών απαγωγών μόνο, τίθεται το θέμα. Και στις περιπτώσεις αυτές η βούληση του ανήλικου έχει μια πολύ συγκεκριμένη αξία σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση. Τώρα αν δούμε την επόμενη διαφάνεια βλέπουμε η θέληση του ανήλικου οδηγεί σε πολύ συγκεκριμένες συνέπειες. Εφόσον υπάρξει σωστή ακρόαση δημιουργείται μια κατάσταση όπου μια απόφαση η οποία λαμβάνεται σε μια χώρα θα μπορούσε να μην γίνει δεκτή σε μια άλλη χώρα και έχουμε να κάνουμε τότε με ε, διαφορετικού με ε, μη αναγνώριση των αποφάσεων μιας χώρας στις υπόλοιπες. Βλέπουμε επίσης και το αντίθετο, ότι όταν κάποιος, ένας ανήλικος περνάει από μια ακρόαση η οποία θεωρείται σωστή, η διαδικασία κανονικά θα μπορούσε να οδηγήσει στην επιστροφή του ανήλικου. Αυτά είναι κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες είχαμε συζητήσει και στα πλαίσια του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου, του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το θέμα είναι τι θα γίνει στο μέλλον. Από εδώ και πέρα. Θα δούμε ότι η πρόταση την οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2016, έχετε δύο λεπτά, Θα κλείσω λοιπόν λέγοντας, λέει ο μιλητής, ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το τι θα πρέπει να κάνουμε στο μελλοντικό κανονισμό που θα πρέπει να βελτιώσει την κατάσταση, γιατί με τις ισχύουσες διατάξεις τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε ε, δυσκολίες γιατί η ακρόαση και η μαρτυρία ενός ανήλικου σε μια χώρα μπορεί να γίνει αποδεκτή και έγκυρη και σε άλλες χώρες όχι. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την ακρίβεια της παρέμβασής σας. Τελμπερχάιντα Καζνάβα. Είστε στη χωροφυλακή, τη γαλλική χωροφυλακή, αποτροπή ε, εγκληματικών συμπεριφορών ε, των ε, νέων και ανηλίκων και είστε και ε, νομικός και θα μας μιλήσετε για το θέμα της παιδικής ηλικίας σε κίνδυνο. Σας ευχαριστώ με τιμά ιδιαίτερα που μπορώ να συζητήσω μαζί σας μία ημέρα πριν την επέτειο της Διεθνούς Σύμβασης των δικαιωμάτων του Παιδιού. Εργάζομαι εδώ και 20 χρόνια στο θέμα της προστασίας των παιδιών και όπως είπατε και εσύ, ε, έχω δύο ρόλους, όπως συχνά λέω ότι έχω δύο μειονεκτήματα, αστείο είναι σε τέτοιες συναντήσεις όπως ε, σε ημερά ουσιαστικά ε, δικαιολογείται ο γάμος μεταξύ του δικαίου και της ψυχολογίας ε, και μπορώ να πω ότι κύριε Φορκάτα Μιράντα χάρηκα πολύ που σας άκουσα και νομίζω ότι και η δική μου παρέμβαση θα είναι συμπληρωματική στη δική σας. Θα το κρίνετε εσείς για να προσεγγίσουμε τώρα το θέμα της ακρόασης ε, των παιδιών ε, στην περίπτωση που έχουμε διεθνείς ε, μάλλον διασυνοριακές οικογενικές διαφορές αυτό μπορούμε να το κάνουμε με δύο τρόπους και καθώς έχω μόνο 15 λεπτά στη διάθεσή μου θα ήθελα να σας δώσω κάποια ουσιαστικά μηνύματα μέσω της εμπειρίας μου και μέσω δύο συγκεκριμένων υποθέσεων που αφορούν τους ανηλίκους. Το πρώτο που θέλω να σας πω για να κατανοήσετε αυτή την ε, πρακτική και αφορά στη δουλειά μου είναι ότι ε, το τμήμα του οποίου είμαι επικεφαλής λέγεται τμήμα πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας. Είμαστε πέντε άτομα, είμαστε ε, ειδικοί ε, και εργαζόμαστε στην Ζηρόντ, αλλά και οι πέντε έχουμε καταρτιστεί για την ακρόση των ανηλίκων αυτών. Όλοι είμαστε εθελοντές και όλοι έχουμε εξειδικευτεί στην ακρόση των ανηλίκων. Το δεύτερο που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι ακούμε παιδιά στα πλαίσια δικαστικής διαδικασίας, αλλά αποκλειστικά και στο πλαίσιο της ποινική διαδικασίας και όχι στο πλαίσιο της αστικής διαδικασίας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι όταν ε, ακούμε τα παιδιά, ένας Γάλλος... Ε, δικαστής ε, επιμελείται του θέματος, ε, είτε ένας ε, δικαστής ποινικό, ένας δικαστής για παιδιά ή ένας ανακριτής και αναλαμβάνει την έρευνα ο χωροφύλακας του τμήματος και όταν φτάνουμε στο στάδιο της ακρόασης του ανελίκου, τότε το αναλαμβάνει το δικό τμήμα γιατί είμαστε ειδικοί. Είναι σημαντική λεπτομέρεια αυτή για να κατανοήσετε καλύτερα από πού μιλώ. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά ε, τα οποία ακούμε συχνά είτε είναι θύματα ε, είτε μάρτυρες ε, σε ένα φάκελο που έχουμε ποινικέ διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Συμπληρωματικά ακούμε τα παιδιά γκρόσο ε, μόντο από τη στιγμή που είναι σε ηλικία να μπορούν ε, να μιλήσουν ε, στο πρώτο ενικό, στο πρώτο πρόσωπο ενικού λέγοντας εγώ δηλαδή και θεωρούν ότι είναι ένα ξεχωριστό άτομο από τη μητέρα και να μπορούν να χειριστούν και ε, το λόγο σε έναν βαθμό. Ε, εγώ, καθώς όπως σας είπα είμαι και ψυχολόγος, ε, αλλά και ανακρίτρια, ο ανακριτής αναζητά την αλήθεια, τουλάχιστον την αντικειμενική εκδοχή των γεγονότων και θα πρέπει το παιδί να μπορεί τουλάχιστον να χειριστεί τη γλώσσα και ε, να μπορούμε να προσαρμοστούμε στις γνωστικές του ικανότητες. Τα πιο μικρά παιδιά λοιπόν ε, από 3 ως 12 ε, ετών ακούμε και επίσης και τους ανηλίκους που έχουν ε, πολύπλοκες ε, διαδρομές, ε, μπορεί να παρουσιάζουν κάποιες παθολογίες ή κάποιες αναπηρίες και σε αυτές τις περίπλοκες καταστάσεις βρίσκουμε παιδιά που ενέχονται σε διάφορες διασυνοριακές διαφορές μεταξύ των γονιών και μπορεί να έχουν έρθει βία στην Γαλλία και ε, ακόμη και αν ένας γονιός ε, είναι Γάλλος, μπορεί να μην μιλούν γαλλικά ή να μιλούν κακά γαλλικά. Έτσι λοιπόν, ε, έρχομαστε εμεί εδώ συμπειρογνώμονε. Θα σας ε, εξηγήσω την πρακτική μου και θα μου πείτε αν ορθή ή όχι. Πάντω είναι σημαντικό να επενθυμίσω ότι τα παιδιά για πολύ καιρό στη Γαλλία δεν ακούγονταν. Τιμολογικώ μιλώντα το παιδί έρχεται όρος ε, από το infants, από τα λατινικά και αυτό σημαίνει αυτός που δεν μιλά. Και οι Γάλλοι δικαστές για καιρό θεωρούσαν ότι δεν ήταν πολύ σημαντικό να ακούνε τα παιδιά γιατί είτε θεωρούσαν ότι τα παιδιά έλεγαν πολλά ψέματα είτε ότι δεν ήταν ικανά με τη μη ε, νομική έννοια του όρου, δηλαδή ότι δεν ήταν πολύ σημαντικό να έχουμε ακρόση των παιδιών αυτών. Όμως, εδώ και κάποιο καιρό τώρα, ε, εγώ εδώ και 20 χρόνια που σας επασχολούμαι με το θέμα αυτό ε, και από το 1998 ακούμε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον το τι έχουν να πούν τα παιδιά και το σημαντικό είναι ότι όχι απλώς ακούμε τα παιδιά, αλλά προσπαθούμε να συμφιλιώσουμε και τα λόγια των παιδιών με ε, την ευημερία τους, αλλά και με τα τραύματα που μπορεί να έχουν βιώσει. Γι' αυτό σας ε, έφερα ε, δύο περιπτώσεις με τις οποίες ασχολούμαστε στον Πορντό. Λοιπόν, τώρα το πρώτο παράδειγμα είναι η καταγγελία από έναν από τις δύο γονείς κατά ε, του άλλου ε, για βίαιη συμπεριφορά ή επίθεση σεξουαλική ε, κατά ενός ή περισσότερων παιδιών του ζευγαριού. Η πρώτη δυσκολία είναι να ανακαλύψουμε ποια είναι η αλήθεια, να αναδειθεί η αλήθεια. Είναι πάρα πολύ πολύπλοκο αυτό αν δεν υπάρχουν αποδείξεις, γιατί έχουμε το λόγο του ενός έναντι του άλλου. Και όταν η φάκελη είναι εσωτερική, οι παθέσεις είναι εσωτερικές στην Γαλλία, ήδη είναι ε, πολύπλοκο. Αλλά όταν ε, έχουμε και ε, ένα εξοδαφικό στοιχείο στη διαδικασία, καταλαβαίνετε ότι γίνεται πάρα πολύ πολύπλοκο για την έρευνα. Έτσι λοιπόν τώρα η ερώτηση που θέτω εγώ με το δικό μου ρόλο είναι για ποια αλήθεια μιλάμε. Αν ε, μιλήσουμε από τη σκοπιά του νομικού η αλήθεια είναι περισσότερο η ιστορική δικαστική αλήθεια, δηλαδή η αντικειμενική αλήθεια των γεγονότων, ενώ αν μιλήσω ως ψυχολόγος ε, τότε μιλάμε για την υποκειμενική αλήθεια περισσότερο, δηλαδή την αλήθεια του υποκειμένου. Πώς συμφιλιώνουμε τα δύο γνωρίζοντας ότι αυτά δεν επικαλύπτονται παρτίτως σε τέτοιε υποθέσει, ε, εμεί επαγγελματίε πρέπει να έχουμε δύο υποθέσει εργασία. Η πρώτη είναι ότι ε, αν αυτό που θα καταγγείλουν οι γονείς ε, είναι αλήθεια, δηλαδή αν ισχύουν οι βιοπραγίες ή οι σεξουαλικές επιθέσεις κατά του παιδιού ή αν πρόκειται για μια ψευδή καταγγελία ε, και ο γονέας ε, που κατηγορείται δεν έχει διαπράξει αξιόπινες πράξεις και δεν υπάρχει κακομεταχείριση του παιδιού. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι έχει χρησιμοποιηθεί το παιδί από τον γονέα που ε, κάνει την καταγγελία και πολύ συχνά είναι όμοιρος το παιδί. Οι συνέπειες για τα παιδιά αυτά είναι πάρα πολύ βαριές. Ο ψυχίατρος Γκάρνεν έχει μιλήσει για σύνδρομο γονικής αποξένωσης. Είναι πολεμικός όρος και δεν θα αναφερθώ εγώ σε αυτό σήμερα γιατί δεν έχω χρόνο. Αλλά θα προτιμούσα να μιλήσω ε, για επιρροή, άσκηση επιρροή από το γονέα στο παιδί. Αλλά όποια ρολογία και να χρησιμοποιήσουμε, ο μηχανισμό για το παιδί που είναι αντικείμενο χειραγώγηση είναι ο ίδιο. Είναι σημαντικό για μα ε, να πρέπει να, να χωρίσουμε την ήρα από το στάρι. Είναι πολύπλοκο και γι' αυτό ε, βλέπετε ο μύθος της Αριάδνης που θα είναι η κατάρτιση των ε, επαγγελματιών. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη περίπτωση όταν έχουμε ψευδείς καταγγελίες και όπως σας είπα, όταν έχουμε και την εξοδοφικότητα γίνεται ακόμη πιο πολύπλοκο. Τώρα, η δεύτερη περίπτωση που αντιμετωπίζουμε στο τμήμα μου είναι το να ακούμε τα παιδιά σε περίπτωση που έχουμε ενδοοικογενειακή βία ε, και όταν η βία αυτή γίνεται μεταξύ ζευγαριών που κατοικεί αλλού εκτός Γαλλίας ή όταν ο ένας από τους γονείς είναι Γάλλος. Ε, 95% των περιπτώσεων θα πρέπει να ακούσουμε ε, παιδιά που έχουν επιστρέψει στη Γαλλική επικράτεια με τη μητέρα τους. Πολύ συχνά ε, έτσι έχει. Ε, έτσι έχουν οι περιπτώσεις αυτές. Το 2018, σύντομα 2019, εγώ θέλω να δηλώσω ικανοποιημένη που είχε αλλάξει το παράδειγμα στη Γαλλία και ε, πολλές ε, φορές ε, ακούω να μου λένε ότι όταν πρόκειται για παιδιά είναι απλώς μάρτυρες τα παιδιά αυτά της ενδοκογενικής βίας, επομένως δεν χρειάζεται να τα ακούσουμε. Σήμερα και καθημερινά εργάζομαι εκεί λέω και δεν είμαι η μόνη, καθημερινά δηλαδή το δουλεύω αυτό, λέω ότι τα παιδιά που ζουν σε ένα ε, τέτοιο δηλητηριώδες ε, κλίμα ενδοκογενειακής βίας είναι θύματα, είναι θύματα, τα παιδιά είναι θύματα, δεν είναι μόνο μάρτυρες. Ακόμη και αν ε, δεν έχουν δεκτεί προσβολές ή ξύλο, τα παιδιά αυτά είναι θύματα. Έτσι λοιπόν σε αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις αυτό που καθιστά δύσκολη τη δουλειά μας ως ανακριτές είναι ε, οι περιπτώσεις παιδιών ε, που ε, είναι προσκολλημένα στους γονείς, είναι πιστά στους γονείς ε, και ε, πολύ αδέξια θα πρέπει να ρωτήσουμε τα παιδιά που προτιμούν να ζουν, τι συμβαίνει και να θέσουμε στους δικούς τους ώμους το βάρος της επιλογής του δικαστή, δηλαδή για το πού πρέπει να ζήσει αυτό το παιδί, με ποιον πρέπει να τοποθετηθεί, αν θα πρέπει να μείνει στη Γαλλία με τη μητέρα του ή αν θα πρέπει να επιστρέψει στον πατέρα που επίσης ζητά την κυδαιμονία. Τώρα, μπορώ να σας μιλήσω για όρους εργασίας. Μήπως μπορούμε να επανέλθουμε στην προηγούμενη διαφάλεια εδώ βλέπετε, δεν βλέπουμε τέλος πάντων πολύ καλά, δυστυχώς λόγω του φωτός. Εδώ νοργικά θα έπρεπε να δείτε μια αίθουσα υποδοχής, όπου υποδεχόμαστε τα παιδιά που θα έρθουν είτε μόνα τους είτε με συνοδεία. Όταν ε, οι γονείς ε, δεν κρίνεται ότι προστατεύουν επαρκώς τα παιδιά, είναι σημαντικό να μπορέσουμε να υποδεκτούμε αυτά τα, τα παιδιά ε, μέσω με έναν ad hoc administrator ε, ή με έναν δικηγόρο. Είναι σημαντικό βλέπω τρέχει και ο χρόνος. Η δουλειά που κάνουμε με τα παιδιά αυτά στην αίθουσα υποδοχής πριν να περάσουμε στην αίθουσα της ακροματικής διαδικασίας να χρησιμεύσει για να μειώσουμε το άγχος τους, να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη τα συναισθήματά τους και είναι ασταθή πολλές φορές τα συναισθήματά τους. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και αυτά τα αντιφατικά συναισθήματα, το θυμό, το φόβο που νιώθουν, τη λύπη, την αγάπη, την απελπισία, την ενοχή, την τροπή και αυτά τα μοιράζονται όλα τα θύματα ε, σε όλο τον κόσμο. Και μάλιστα πολύ περισσότερο αυτά τα παιδιά στις υποθέσεις ε, που σας παρουσίασα, σε αυτές τις ποινικέ υποθέσεις. Αυτή είναι λοιπόν η αίθουσα ακρόασης. Ε, στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε την αίθουσα της ακρόασης. Όταν μιλάμε για ποινικέ υποθέσεις, ε, έχουμε ε, βιντεοσκόπηση ε, των ακροάσεων γιατί μπορούμε έτσι να εργαστούμε και σε επίπεδο μη προφορικής επικοινωνίας. Στη δεύτερη φωτογραφία βλέπετε το χώρο που καταλαμβάνει το παιδί. Βλέπουμε συνήθως δύο πολυθρόνες και αφήνουμε το παιδί να εγκατασταθεί εκεί είναι πολύ σημαντικό και θα τελειώσω στα δύο λεπτά που μου απομένουν. Είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου ότι δεν είναι ένα ε, ενήλικος μινιατούρα το παιδί. Για να μπορέσουμε να ακούσουμε το παιδί θα πρέπει να είμαστε καταρτισμένοι. Δεν μπορούμε να απευθυνθούμε σε ένα παιδί τριών ετών όπως θα κάναμε ε, σε ένα παιδί 11 ετών ή σε ένα παιδί 17 ετών και θα πρέπει να έχουμε τι ελάχιστε γνώσει για το γνωσιακό ε, στάδιο ανάπτυξης ε, του παιδιού, για το κοινωνικό στάδιο της ανάπτυξης. Θα πρέπει επίσης να γνωρίσουμε τα τραύματα που προκαλούν αυτές ε, οι βιοπραγίες στα παιδιά. Τα παιδιά αυτά είναι όμοιροι μεταξύ των δύο γονιών, βρίσκονται στη μέση και τελικά πρέπει να τους ζητήσουμε να διαλέξουν ουσιαστικά θα πρέπει να ξέρουμε πώς λειτουργεί και αυτή η σύγκρουση για το σε ποιον είναι πιστό το παιδί. Έτσι λοιπόν εγώ εργάζομαι και, με, ε, και στην κατάρτιση των δικαστών στην Εθνική Σχολή ε, Κατάρτισης Δικαστών. Εργάζομαι μαζί με τους επαγγελματίες του κλάδου της υγείας, ε, της παιδείας και τους κοινωνιολόγους. Όλοι οι επαγγελματίες που εργάζονται για την προστασία των ανηλικών θα πρέπει να είναι καταρτισμένοι για να ακούσουν τα παιδιά είτε πρόκειται ε, για δικαστική είτε για εξοδικαστική διαδικασία στην Γαλλία και στη Την καθημερινά. Προσπαθούμε ε, να έχουμε αυτή την, ε, αυτό το πολυτομεακό προφίλ. Θα ήθελα να πω ότι για μένα η κατάρτιση αποτελεί μία από τις λύσεις για την πρόληψη και θα πρέπει να έχουμε φυσικά κατά νου και το διεθνές δίκαιο για την κατάρτιση των εμπειρογνωμένων, αλλά υπάρχει και η κατάρτιση που αφορά την ψυχολογία ε, των παιδιών αυτών. Ε, σίγουρα έχει κόστος η κατάρτιση, αλλά ε, Πρέπει να έχουμε τα μέσα για τη χάραξη πολιτική μα ε, και θεωρώ ότι τα χρήματα που επενδύουμε στην πρόληψη και στην κατάρτιση πάντοτε θα κοστίζουν ε, λιγότερο σε σχέση με τις δαπάνε υγείας και ασφάλειας ε, που προκαλούνται από την διάπραξη βίας. Σα ευχαριστώ που με ακούσατε. Σας ευχαριστούμε για τη μαρτυρία σας που μοιραστήκατε τις πεπιθήσεις σας και την πείρα σας μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και θα ήθελα να σας ευχηθώ και χρόνια πολλά. Γιατί ξέρω και ότι ο σας είναι εδώ στην αίθουσα και σας ακούει. Χρειάζονται λουλούδια, λέει ο πρόεδρος. Να περάσουμε τώρα στο τελευταίο πάνελ που αφορά τώρα την διαμεσολάβηση. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένα για το θέμα αυτό. Για την επίλυση των οικογενειακών διαφορών. Η διαμεσολάβηση θα μπορούσε να οδηγήσει τους γονείς να σκεφτούν εκ νέου τι ευθύνε τους προκειμένου να βρουν από κοινού μακροπρόθεσμε λύσεις για το παιδί τους. Έχουμε τώρα δύο εμπειρογνωμόνε, την κυρία Άλισον Σάλαμπη, η οποία είναι CEO της ε, ε, Reunited International, βρετανική οργάνωση παγκόσμιας φήμης και εξειδικεύεται στην διασυνοριακή διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις απαγωγής παιδιών. Έχουμε, ε, μάλλον ε, το κέντρο ακούει πάνω από 17.000 υποθέσεις ε, και προσφέρει κάθε χρόνο υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε πάνω από 1.000 οικογένειες. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για να μας μιλήσετε για τη διαμεσολάβηση. 15 λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε σήμερα εδώ. Όπως αναφέρατε ήδη, η United είναι μια κυβερνητική οργάνωση που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο υπό την ε, εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών ε, και Δικαιοσύνη. και έχουμε δύο βασικές υπηρεσίες οι οποίες ε, προσφέρουμε. Καταρχήν μια τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης η οποία λαμβάνει ασχολούνται με 500 έως 600 σε περιπτώσεις απαγωγής παιδιών ετησίως και εδώ βέβαια δίνουμε συμβουλές και υποστηρίζουμε τόσο τον Απαγωγή γονέα, και τον γονέα ο οποίος είναι το θέμα αυτής της απαγωγής και έτσι ε, γνωρίζουμε από την πρακτική μας ε, το τι λειτουργεί καλά και το τι δεν λειτουργεί τόσο καλά. Η δεύτερη υπηρεσία που προσφέρουμε είναι ακριβώ η διαμεσολάβηση σε διεθνεί υποθέσει και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τι διεθνεί υποθέσει ακριβώ απαγωγή ε, παιδιών. Όπω είπατε ήδη, η διαμεσολάβηση ακούει το ένα και περισσότερο ω δυνητικό τρόπο επίλυση τέτοιων υποθέσεων. Ωστόσο, πολύ λίγες υποθέσεις ε, τέτοιου είδους ε, δηλαδή απαγωγέ ε, παιδιών προχωρούν στη διαμεσολάβηση. Εμείς ξεκινήσαμε από το 2001 με αυτή την υπηρεσία και από το, έως το 2014 διαπιστώσαμε ότι οι σχετικές είχαν μειωθεί ε, σημαντικά στον διαμεσοδιάστημα. Δηλαδή οι γονεί δεν γνώριζαν ότι υπάρχει διαμεσολάβηση και αρμόδιοι ε, νομικοί ε, και οι επαγγελματίε του χώρου δεν του ενημέρωναν για αυτή τη δυνατότητα και αντιθέτω του αποθάρρυναν κιόλα. Άρα λοιπόν εμεί απευθυνθήκαμε στην αρμόδια υπηρεσία και είπαμε ότι θέλουμε να εισαγάγουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα διαμεσολάβηση και να περάσουμε λίγο στην προηγούμενη διαφάνεια. Ε, και τι θα σήμαινε αυτό, ότι θα υπάρχει ένας ε, διαμεσολαβητής ε, παρόντας στο αρμόδιο δικαστήριο, δηλαδή δικαστήριο το οποίο εκδικάζει όλες τις σχετικές υποθέσεις, είτε εντάσσονται στη Σύμβαση της Χάρης είτε όχι. Έτσι λοιπόν το αρμόδιο Υπουργείο ενέκρινε αυτό το σύστημα και δόθηκαν κάποιες κατευθυντήρες γραμμές για τους επαγγελματίε ω προ το πώ να διαχειρίζονται αυτέ τι υποθέσει, αλλά και αναλύοντας πώς σε κάθε υπόθεση στο πλαίσιο αυτού του πιλωτικού προγράμματος ε, θα ε, ενθαρρύνονταν οι γονείς να αξιοποιήσουν τον διαμεσολαβητή. Αυτό που ισχύει εδώ είναι ότι έχει εθελοντικό χαρακτήρα διαμεσολάβηση. Ο δικαστής δηλαδή δεν μπορεί να επιβάλλει τη διαμεσολάβηση, μπορεί μόνο να την ενθαρρύνει. Ε, ε, τον Μάρτιο λοιπόν τώρα του 2018 είχαμε τα αποτελέσματα ή μάλλον συγγνώμη ξεκίνησε ε, το πρόγραμμα από τον Απρίλιο συγκεκριμένα εγκρίθηκε τον Μάρτιο και εγκρίθηκε τον Απρίλιο και βλέπουμε ε, εδώ στην επόμενη διαφάνεια ότι όταν ξεκίνησαν αυτές οι κατευθυντήρες γραμμές είχαμε μία, ένα άμεσο αντίκτυπο Δηλαδή το 2018 είναι με πράσινο χρώμα και σε κόκκινο χρώμα το 2017. Βλέπετε πόσο αυξήθηκαν λοιπόν άμεσα οι ε, σχετικέ παραπομπές για διαμεσολάβηση λόγω ακριβώ των κατευθυντηρογραμμών. Και στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε τον αριθμό των υποθέσεων για τι οποίε έγινε διαμεσολάβηση. Και για μία ακόμα φορά βλέπουμε πω οι υποθέσεις εκείνες οι οποίε παραπέμφθηκαν στη διαμεσολάβηση ε, αυξήθηκαν σε ό,τι αφορά τον αριθμό του στο πλαίσιο του, ε, που έτρεξε το πιλωτικό πρόγραμμα και διαπιστώσαμε ότι στο 66% των περιπτώσεων που παραπέμφθηκαν σε διαμεσολάβηση κατάφεραν να καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα. Εδώ δηλαδή οι ε, γονείς έρχονται σε διαμεσολάβηση ε, για 9 ώρες σε διαχρονικό διάστημα 2 ημερών και σε αυτές τις 66 λοιπόν ε, περιπτώσεων δεν χρειάστηκε να υπάρξει εκδίκαση της υπόθεσης. Έγινε δηλαδή φιλικά ο διακανονισμός. Άρα λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που θα πρέπει να πληρούνται ως προϋποθέσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει η διαμεσολάβηση. Καταρχήν, υποστήριξη από την πλευρά των δικαστών. Αλλά δεν μόνο η υποστήριξη των δικαστών, είναι και η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού νομικού συστήματος και νομικής διαδικασίας σε συγκεκριμένη χώρα. Εάν δούμε δηλαδή ε, αυτές τις περιπτώσεις της Χάγης, όπου δηλαδή ένας ε, γονέας ε, θα απαγάγει ένα παιδί επειδή ο άλλος γονέας δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, γνωρίζουμε πως η διαμεσολάβηση δεν θα λειτουργήσει γιατί ξέρουμε ότι αυτός ο γονέας ε, γνωρίζει ότι θα τρέξει το, η διαμεσολάβηση για ένα, δύο, τρία χρόνια και αυτό δεν τον συμφέρει γιατί μετά από αυτό το περίοδο, περίοδο μπορεί να εκδοθεί η απόφαση με βάση την οποία πράγματι η κατακράτηση του παιδιού έγινε παρανόμως αλλά μέσα σε αυτή την περίοδο έχει προσαρμοστεί το παιδί στη νέα πραγματικότητα. Άρα λοιπόν ποιο είναι το κίνητρο για να ε, προτιμήσει τη διαμεσολάβηση. Δεν υπάρχει. Ε, μία ακόμα απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποστήριξη των νομικών επαγγελμάτων και στην Ηνωμένο Βασίλειο αυτό είναι και το βασικό πρόβλημα. Αυτή είναι η βασική πρόκληση γιατί εδώ θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία ε, των ε, νομικών, των επαγγελματιών του κλάδου γιατί η ενστικτόδης αντίδραση αν θέλετε ενός δικηγόρου είναι ακριβώς να προτιμήσει την δικαστική λύση. Για αυτούς δηλαδή αποτελεί νομικό πρόβλημα το οποίο χρήζει νομικής λύσης. Άρα λοιπόν υπάρχει μια διάσταση απόψεων αν θέλετε σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίε από το χώρο ε, του δικαίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ίμιση δηλαδή υποστηρίζει τη διαμεσολάβηση ως εργαλείο, ενώ το άλλο ίμιση είναι εχθρικό απέναντι στη διαμεσολάβηση, ενώ κάποιοι γονείς με τους οποίους μιλήσαμε ε, μας είπαν ότι οι δικηγόροι τους τους αποθαρρύνουν, γιατί θεωρούν ότι ε, και θα καθυστερήσει όλη η διαδικασία και το αποτέλεσμα δεν θα είναι πολύ καλό. Άρα λοιπόν αυτή είναι τεράστια πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Το πλεονέκτημα ωστόσο που έχουμε είναι ότι υπάρχει νομική συνδρομή για όλους τους ενάγοντες γονείς στο πλαίσιο της Σύμβασης της Χάγης με βάση την οποία καλύπτονται τα έξοδα ε, για την ε, ε, διαμεσολάβηση. Δηλαδή ο ενάγων γονέας δεν ε, καταβάλει έξοδα και υπάρχει και χρηματοδοτική υποστήριξη προκειμένου να μεταβεί ο ενάγων γονέα σε άλλο κράτο μέλο για να συμμετάσχει στη διαμεσολάβηση. Και εδώ δηλαδή αναφέρομαι και στην πτήση αυτού του γονέα όσο και στο κόστο τη διανεκτέρευση των διανεκτέρευσεων. Και αυτό το λέμε γιατί ε, θεωρούμε και διαπιστώσαμε ότι πάντοτε είναι καλύτερο οι γονεί να βρίσκονται παρόντε στην ίδια αίθουσα και να κάθονται και να συζητούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Επίσης υπάρχει και μια νομική αρρωγή για τον εναγόμενο γονέα σε ό,τι αφορά ε, τον, τις δυνατότητες ε, που έχει και κατά πόσο μπορεί να λάβει τέτοια υποστήριξη. Και στο ίμιση των περιπτώσεων πράγματι λαμβάνει αυτή την υποστήριξη. Δηλαδή το ίμιση των εναγόμενων γονέων λαμβάνει από την κάλυψη των εξόδων του. Και ακόμα και αν δεν εγκριθεί υπάρχει και ένα ε, περαιτέρω υποστηρικτικό πρόγραμμα γιατί ε, θεωρούμε πως χρημα... προβλήματα οικονομικής φύσης δεν θα πρέπει να αποτελέσουν κόλλημα προκειμένου ένας γονέας να μπορέσει να συμμετάσχει σε μια διαδικασία διαμεσολάβησης. Κάτι ακόμα που θεωρούμε ως χρήσιμο είναι η ε, διαμεσολάβηση μέσω του διαδικτύου. Δηλαδή μπορούμε να αξιοποιήσουμε το Skype ή το Zoom για να το κάνουμε. Προτιμούμε βέβαια οι γονεί να μεταβαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, και να είναι παρόντε για τη διαμεσολάβηση, αλλά αν δεν μπορούν να το κάνουν, γιατί για παράδειγμα ένα γονέο βρίσκεται στη Νέα Ζηλανδία ή στην Αυστραλία, δεν μπορεί να λάβει για παράδειγμα γέρο τη θεώρησή του, τότε μπορεί να γίνει διαμεσολάβηση μέσω Skype. Και ναι, στέφεται με επιτυχία, αλλά δεν είναι τόσο αποτελεσματικό ως εργαλείο σε σύγκριση με τη φυσική παρουσία των ε, γονέων για να υπάρξει και πάλι επικοινωνία μεταξύ τους, να αποκατασταθεί επικοινωνία μεταξύ τους. Κάτι ακόμα που μας ανησυχούσε ε, στη διαμεσολάβηση ήταν ότι οι γονείς ε, προσέρχονται στη διαμεσολάβηση, συζητούν, φτάνουν σε μια συμφωνία ε, και μετά χωρίζονται. Εμείς όμως δεν γνωρίζουμε τελικά τι έγινε με αυτή τη συμφωνία. Αξιοποιήθηκε σωστά, είχε βάθος χρόνου, ήταν βιώσιμη ή για παράδειγμα δεν λειτουργήσε για πολύ χρόνο και τελικά προσέφυγαν στην ε, δικαστική λύση. Και έτσι λοιπόν ήρθαμε σε επαφή με γονεί ε, του οποίους ε, είχαμε προσφέρει διαμεσολάβηση πριν από 6, 7, 8 χρόνια ναι, και σε όλε τι περιπτώσει στι οποίε λοιπόν απευθυνθήκαμε σε αυτού του γονεί, με μεγάλη μα χαρά διαπιστώσαμε ότι αυτή η συμφωνία είχε αντέξει ε, ε, στο χρόνο. Δηλαδή δεν χρειάστηκε να, να θεωρήσει κανένα γονέα αυτή τη συμφωνία και με βάση του όρου τη συμφωνία ε, συνεχιζόταν αυτή η συμφωνία καθώ όλοι είχαν συμφωνήσει. Ε, και με αυτόν τον τρόπο είχαν τη δυνατότητα και τα παιδιά σε αυτές τις υποθέσεις να διατηρήσουν μία ε, ουσιαστική σχέση και με τους δύο κονείς. Ποια είναι λοιπόν τα εμπόδια σε ό,τι αφορά ε, την, ε, για τη διαμεσολάβηση είναι ακριβώς ε, η, το αντίθετο από εκείνα που μπορούν να βοηθήσουν από τα πλεονεκτήματα, δηλαδή ελλειπής υποστήριξη από τους δικαστές και γενικότερα από τους επαγγελματίες του χώρου, γιατί θεωρούν ότι ακριβώς πρόκειται για νομικό πρόβλημα που χρήζει νομικής λύσης. Επίσης υπάρχει και το ζήτημα της ελλειπούς ευαισθητοποίησης τη κοινή νόμης. Δηλαδή πολλοί γονεί και στον Ηνωμένο Βασίλειο και γενικότερα στην ε- Ευρώπη δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα της διαμεσολάβησης. Ε, και τέλος ένα τεράστιο ε, εμπόδιο είναι ότι δεν υπάρχει σε πολλά κράτη-μέλη οικονομική υποστήριξη για τη συμμετοχή στη διαμεσολάβηση και αυτό αποτελεί μια μεγάλη ανησυχία για πολλούς γονείς οι οποίοι δηλαδή βρίσκονται σε μια τέτοια διαδικασία εντός, εκτός συγγνώμη, Ηνωμένου Βασιλείου και ε, θεωρούν τις βάστα αυτό το κόστος. Άρα λοιπόν το πιλωτικό πρόγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2019, ε, καθώς ξεκίνησε τώρα τον Απρίλιο του 2018, αλλά ήδη έχουμε σε, σε ε, επαφή με τους αρμοδίους δικαστές για να υπάρξει μια παράταση κατά ένα χρόνο, γιατί όπως σας είπα χρειάζεται να λάβει η χώρα μια αλλαγή νοοτροπίας και ε, δεν μπορούμε να επιτύχουμε μια τέτοια αλλαγή νοοτροπίας σε ένα χρόνο και μόνο. Χρειαζόμαστε λοιπόν περαιτέρω χρόνο. Αυτά λοιπόν είναι τα πορίσματα μας με βάση την εμπειρία που έχουμε από τη διαμεσολάβηση. Ε, είναι χρήσιμη, μπορεί να βοηθήσει, δεν είναι ε, βέβαια η κατάλληλη λύση για όλες τις υποθέσεις. Απορρίπτουμε δηλαδή τόσες υποθέσεις ε, στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης όσες ε, αποδεχόμαστε. Αλλά πραγματικά αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο. Σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ κύριε Σέλαμπη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται με τους γονείς οι οποίοι προσφεύγουν στη διαιτησία, στη διαμεσολάβηση. Είναι δεκτική εκ των προτέρων σε αυτού του τύπου διάλογο. Μήπως αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει τα επίπεδα ικανοποίησης, γιατί επιτυγχάνεται ε, στις 60% των περιπτώσεων ή έχουμε να κάνουμε με έναν ετερογενή πληθυσμό ο οποίος προσωμιάζει με το σύνολο της οικογένειας. Νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να δώσουμε απάντηση. Έχει μεγάλη σημασία αν θέλουμε να προωθήσουμε τη διαμεσολάβηση θα πρέπει να γνωρίσουμε σε ποιου είδους γονείς και τις τι νοοτροπίες και αντιλήψεις ανταποκρίνεται. Ο τελευταίος εμπειρογνώμων για σήμερα είναι η κυρία Καλαμιούσομ Είστε δικηγόρος οικογενειακό δίκαιο, ειδικευμένοι σε θέματα διατησίας, σε διασυνοριακές οικογενειακές διαφορές. Είστε και εκπαιδεύτρια. Ε, είσαστε υπεύθυνοι ε, στην υπηρεσία ΜΙΚ, στην οργάνωση ΜΙΚ μάλλον. μία από τις πιο δραστήριες οργανώσεις στον τομέα διεθνών διαμεσολαβήσεων, στον τομέα των οικογενειακών συμβούλων και στα θέματα των οικογενειακών απαγωγών με έδρα του Βερολίνου. Έχετε και εσείς 15 λεπτά στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας και την κυρία Μωρέν Σαρτιέ που μου προσεκάλεσε εξ ονόματος του ΜΙΚ του Διεθνούς Κέντρου Διαμεσολάβησης για Οικογενειακές Συγκρούσεις και Απαγωγές. Η Άλισον είπε προηγουμένως ότι η διαμεσολάβηση δεν είναι κατάλληλη για όλες τις περιπτώσεις. Υπάρχουν γονείς ε, οι οποίοι είναι τόσο, σε τόσο μεγάλο επίπεδο αντιπαράθεσης που είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν σε ένα δωμάτιο και να συζητήσουν αλλά είναι η σωστή επιλογή για αυτούς τους γονείς και εδώ νομίζω αναφέρουμε στην πλειοψηφία των γονέων οι οποίοι έχουν κατανοήσει ότι είναι προς όφελος του παιδιού τους, της ευτυχίας τους, της ευημερίας του παιδιού τους να προσπαθήσουν να λύσουν τη διαφορά τους φιλικά. Οι γονείς αυτοί κατανοούν ότι η ικανότητά τους να διαχειρίζονται τη γονεϊκή τους ιδιότητα για τα επόμενα χρόνια εξαρτάται από τον τρόπο τον σωστό με τον οποίο ακολουθούν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Ενώ ο δρόμος της δικαστικής αποκλειστικά αντιμετώπισης αυξάνει την εχθρότητα ανάμεσα στους γονείς εις βάρος των δικαιωμάτων των παιδιών. Εγώ θα αναφερθώ σε προσωπικό επίπεδο ως δικηγόρος σε περιπτώσεις διεθνών διαζυγίων και διεθνών απαγωγών βλέπω ότι όταν έχουν δυσκολίες οι γονείς να διαχειρίζονται τη γωνιακή τους ιδιότητα πριν ξεκινήσουν τις διαδικασίες αυτές, τότε μετά από μακρές δικαστικές διαδικασίες υπάρχουν ε, ελάχιστα πλέον μικρότερα ή λιγότερα περιθώρια. Υπάρχουν συνεχώς αντιπαραθέσεις νομικές που δεν διευκολύνουν την διαδικασία. Πάντως προσπαθούμε να πείσουμε τους γονείς να δουν κυρίως τα συμφέροντα των παιδιών τους. Πολλές φορές τα παιδιά τους τα αγνοούν στα πλαίσια του αγώνα για την κυδαιμονία. Ενώ θα πρέπει να συνεργαστούν για τα παιδιά. Η διαμεσολάβηση είναι κάτι το διαφορετικό από τις δικαστικές διαδικασίες. Εδώ έχουμε έτσι γελιός τον ορισμό. Είναι μια ε, διαφρομένη διαδικασία η οποία περνά μέσα από συγκεκριμένες φάσεις σε εντελώς εθελοντικό επίπεδο και κάθε ε, συνεδρία κρατάει γύρω στις 10 με 15 ώρες. Είναι φυσικά κάτι το ε, απόρριτο και οι διαμεσολαβητές λειτουργούν με τη μέγιστη αντικειμενικότητα τα ωφέλη για τους γονείς είναι σαφή και τεκμηριωμένα. Στη μελέτη αξιολόγησης του 2015 υποθήκε ότι η διαμεσολάβηση είναι και πιο αποτελεσματική και πιο ταχεία από τις δικαστικές διαδικασίες. Αυτό οφείλεται στο ότι οι ίδιοι οι γονείς είναι οι ίδιοι αρχιτέκτονες της συμφωνίας. Πρόκειται για αναγνώριση των δυνακοτήτων τους και στήριξη της διαδικασίας. Η διαμεσολάβηση οδηγεί τους γονείς να κατανοούν ότι δεν είναι πλέον ζεύγος, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουν να συνεργάζονται ως γονείς. Ε, προσπαθούμε να αλλάξουμε τις αντιλήψεις των γονέων και οι διαμεσολαβητές χρησιμοποιούν μέσα και τεχνικές για να το πετύχουν. Σαν παράδειγμα, το να ζητάμε στα παιδιά στα πλαίσια μιας διαμεσολάβησης το πώς ε, θα βλέπουν τα παιδιά τους αυτή την υπόθεση μετά από 10-15 χρόνια. Πώς θα βλέπουν με μάτια ενήλικα τις διαδικασίες αυτές. Είναι μια σκληρή ερώτηση η οποία κάνει τους γονείς ίσως ε, να το δουν διαφορετικά. Η έρευνα δείχνει ότι δεν είναι ο χωρισμός ε, που δημιουργεί προβλήματα στα παιδιά, αλλά ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο χωρισμός όταν υπάρχουν διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές σε διαφορετικές χώρες, σε διαφορετικές περιοχές, με διαφορετικές, σε διαφορετικές ζώνες ώρας, όλα αυτά επιβαρύνουν την κατάσταση. Έχουμε περιπτώσεις οι οποίες φτάνουν είτε με email είτε με Skype από πολλές χώρες στον κόσμο είναι δωρεάν και ε, λειτουργούμε σε αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά, πολωνικά, ισπανικά και ιταλικά. Το ΜΙΚ πέρυσι πήρε 213 αιτήματα, έχουμε περάσει για φέτος τους 200 περιπτώσεις, ε, είχαμε εμπλακεί με 65 χώρες, οι περισσότερες χώρες της Ένωσης είναι παρούσες Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις οικογενειακών διαφορών. Ε, κάποιες ε, περιπτώσεις ήταν σύμφωνα με την Συμφωνία της Χάγης, κάποιες άλλες εκτός Χάγης και κάποιες ήταν πρόληψη μετακίνησης. Ε, προσπαθήσαμε εμείς να έχουμε στη διάθεσή μας σωστά εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές, ε, πολύγλωσσους. Έχουμε και άλλες οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα αυτά, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία. Οι διαμεσολαβήσεις αυτές είναι δύσκολες βέβαια και για τους γονείς και για τους διαμεσολαβητές. Οι συγκρούσεις πολλές φορές είναι υψηλής έντασης ε, πολλές φορές οι γονείς έχουν έρθει από το εξωτερικό λίγες μέρες πριν και η διαφορετική γλώσσα και οι διαφορετικές αντιλήψεις πολλές φορές δυσκολεύουν την κατάσταση. Το θέμα είναι η επικοινωνία βέβαια. Ε, και διαχείριση της σύγκρουσης έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε σωστά τη συγκρουσιακή συμπεριφορά όπως επίσης και την δυνατότητα επικοινωνίας στις γλώσσες των γονέων, έστω και σποραδικά. Όταν ένας γονιός θέλει να μιλήσει τη μητρική του γλώσσα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, λόγω του υψηλού στρες πρέπει να γίνεται κατανοητός. το 4B, το μέσο αυτό ε, συνδιαμεσολάβησης, οι διαμεσολαβητές είναι δίγλωση στο μέγιστο δυνατό βαθμό, είναι διαπολιτισμικής προέλευσης και είναι επίσης και διεπαγγελματική, διατομεακή έτσι ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών. Ε, η διάσκεψη της Χάγης δίνει τις κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση των διεθνών απαγωγών. Το ΜΙΚ έχει 150 εξειδικευμένους διαμεσολαβητέ σε 27 χώρες και σε 30 γλώσσες. Όλοι οι διαμεσολαβητές έχουν κάνει ε, την επίσημη διαδικασία κατάρτισης ε, που γίνεται σε αιτήσια βάση ε, στην Γερμανία, στη Σιγκαπούρη και στην Ιαπωνία. Η εκπαίδευση επιτρέπει στους διαμεσολαβητές να συμμετέχουν στους καταλόγους του ΜΙΚ και της Διεθνούς Ένωσης Διαμεσολαβητών ε, στην οποία ανήκουμε και προέρχονται από 11 διαφορετικές χώρες. Ε, το ΜΙΚ και το ΕΚΟ οργανώνουν ένα σεμινάριο κατάρτισης ε, σε συνεργασία με το Missing Center of Europe σχετικά με τα αναγνωρισμένα πλεονεκτήματα τώρα της διαμεσολάβησης για, την, για τον σεβασμό των δικαιωμάτων των παιδιών στη μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρονται στη δραστηριότητά μας στο λεγόμενο παράδοξο της διαμεσολάβησης Πολλές φορές το οικονομικό είναι ένα πρόβλημα. Πολλοί γονείς θέλουν να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση αλλά δεν έχουν χρήματα. Η κεντρική διοίκηση που συνεργάζεται με το ΜΙΚ προβλέπει ε, την χρηματοδότηση της διαδικασίας σε περιπτώσεις κυρίως απαγωγής, αλλά όχι για όλες τις περιπτώσεις. Η έλλειψη γνώσης για τη διαμεσολάβηση είναι και αυτός ένα σημαντικός λόγος. Οι γονείς μας λέγουν ότι καλό θα ήταν να ήξεραν από αυτά πριν ξεκινήσουν τη διαδικασία τη νομική. Πάρει πολλοί δικηγόροι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η διαμεσολάβηση είναι απλή διαδικασία χορήγησης συμβουλών. Συνεπώς λοιπόν υπάρχει ένας δισταγμός, πάρα πολύ λίγοι νομικοί όμως παραπέμπουν, δικηγόροι παραπέμπουν. Πολλές φορές οι δικηγόροι που παραπέμπουν είναι οι ίδιοι διαμεσολαβητές και γνωρίζουν ότι θα παραμείνουν εμπλεκόμενοι καθ' όλη τη διάρκεια της διαμεσολάβησης. Εμείς συστήνουμε στους γονείς να μιλήσουν σε δικηγόρους έτσι ώστε να ξεκινήσουν τις διαδικασίες διαμεσολάβησης ενημερωμένοι. Ελέγχουν γενικά τις διαδικασίες από τις οποίες θα διέλθουν και υπογράφουν επίσης και ένα μνημόνιο κατανόησης το οποίο πρέπει να αναγνωρίζεται και να επικυρώνεται και στις δύο χώρες. Έτσι πολλοί νομικοί και δικηγόροι θα πρέπει να εκπαιδεύονται να αναγνωρίζουν αυτή την πραγματικότητα της διαμεσολάβησης Υπήρξαν κάποια σχέδια προγράμματα εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση των απαγωγών στην Ευρώπη που οδήγησαν και σε μια μεγάλη συνάντηση τον προηγούμενο Ιανουάριο. Οι δικαστές επίσης είναι και αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να αναφέρονται στα θέματα, να παραπέμπουν στα θέ, στις δυνατότητες της διαμεσολάβησης και αυτό φαίνεται και στην ε, οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρόταση για την αναδιατύπωση τώρα των Βρυξελών 2α θα πρέπει να ακολουθήσει τη σωστή κατεύθυνση. Θα πρέπει να γίνεται αναφορά από πλευρά των δικαστικών διαδικασιών, εκτός και αν καθυστερεί τις διαδικασίες αυτές. Στις περιπτώσεις της Χάγης, των περιπτώσεων που εμπλέκονται με τις ρυθμίσεις της Χάγης, λειτουργεί, θα έλεγα, ανασχετικά ε, σε σχέση με την δυνατότητα χρήσης της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Προβλέπονται ε, δύο συναντήσεις ε, που απέχουν μεταξύ τους 10 μέρες. Ο διαμεσολαβητής είναι παρόν στην πρώτη συνάντηση, ενημερώνει και εφόσον οι γονείς ξεκινούν τη διαδικασία δύο-τρεις μέρες μετά. Εμείς προωθούμε το μοντέλο αυτό και στην συνάντηση που γίνεται δύο φορές το χρόνο στα πλαίσια της διαδικασίας της Χάγης. Σαν αποτέλεσμα, πολλοί δικαστές ταξιδεύουν στην Γερμανία και εκπαιδεύονται σε σχέση με αυτά. Η, τα ποσοστά επιτυχίας είναι πολλά υποσχόμενα και στις απαγωγές το 2015 67% επιτυχία, το 2016 90% και το 17 83%. Ένας άλλος τομέας ο οποίος ενδιαφέρει το ΜΙΚ είναι η αναγνώριση ε, των συμπεφωνημένων αποφάσεων τα λεγόμενα package agreements στις διάφορες χώρες. Τα πακέτα αυτά, τα οποία περιλαμβάνουν πολλά θέματα όπως την γονική ευθύνη, οικονομική κάλυψη εξόδων και κτλ. θα πρέπει να προωθούνται διότι εξυπηρετούν τα συμφέροντα των παιδιών και αποτρέπουν τις δικαστικές προσφυγές. Όμως οι δικαιοδοσίες στον τομέα των απαγωγών είναι περίπλοκες και η εφαρμογή αυτών των συμφωνιών πακέτων είναι περίπλοκη και αβέβαιη. Κανένα από τα υπάρχοντα κοινωνικά, κοινοτικά μέσα δεν παρέχουν τις οδηγίες για τη σωστή επιβολή αυτών των αποφάσεων πακέτων, κάτι το οποίο συνιστά μια επιπλέον τροχοπέδη στην εφαρμογή τους. αν υπήρχε η δυνατότητα εφαρμογής σωστότερη ε, θα υπήρχε και αύξηση των προσφυγών στις διαμεσολαβήσεις. Το ΜΙΚ έχει επίσης οργανώσει ένα νέο πρόγραμμα, ένα νοδικό χάρτη που συνδράμει στην, στην εφαρμογή και στην επιβολή, αν θέλετε, ε, των πακέτων συμφωνίας. Τώρα, ε, στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν χώρες ε, χωρίς ε, δυνατότητα επιβολής των προβλεπόμενων από την Σύμβαση της Χάγης, Μέση Ανατολή σαν παράδειγμα, οι περισσότερες χώρες της Μέσης Ανατολής εκτός από το Μαρόκο και την Τουρκία, σε αυτές τις περιπτώσεις η επαφή με το παιδί είναι σποραδική, γίνεται απλά τηλεφωνικά ή σταματάει μετά την απαγωγή. Η διαμεσολάβηση είναι ο μοναδικός τρόπος για να υπάρξει επικοινωνία ανάμεσα στον γονιό που έχει μείνει μόνος του και στο παιδί. Στην ίδια περιοχή αυτή, την περιοχή Μένα, Υπάρχουν διαδικασίες διαμεσολάβησης, εκτιμάται και θεωρείται κάτι το απαραίτητο για να επιλύονται οι διαφορές. Ε, το ΜΙΚ πέρυσι μπορέσαμε να κάνουμε κάποιες αναλύσεις και να συγκαλέσουμε μία συνάντηση εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες ήταν ε, διαπολιτισμικής προέλευσης ε, και ε, φυσικά ομιλούσαν τουρκική και αραβική ανάλογα και μπορέσαμε να καταλήξουμε σε κάποιες οδηγίες για ένα πρόγραμμα διαμεσολάβησης το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει σύντομα. Έχουμε προσκληθεί στο Μαρόκο επίσης για αντίστοιχες τέτοιες καταρτήσεις. Και τέλος έχουμε ένα όραμα μαζί με όλους τους εμπλεκομένους στον τομέα της διαμεσολάβησης. Η διαμεσολάβηση θα πρέπει να γίνει η προτιμόμενη και ε, οικονομικά αντιμετωπίσιμη μέθοδος, έτσι ώστε τα συμφέροντα των παιδιών να προστατευθούν καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλους ε, τους ομιλητές του δεύτερου και του τρίτου πάνελ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις ή αντιδράσεις στην αίθουσα. Εσείς, Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχηθώ όλοι οι νομοθέτες που σχετίζονται με το θέμα των παιδιών να μπορέσουν να, ακούσουν αυτή την εξαιρετική ακρόαστρα, εξαιρετική πραγματικά και σας ευχαριστώ ειλικρινά. Δεύτερον, αν ε, κάποιος από τους ε, συναδέλφους θέλει το λόγο, θα σας δώσουμε λίγα λεπτά. Κύριε Περζερόν, κύριος Μαρίνιο Πίντο, εγώ θέλω να πάρω το λόγο, αλλά ήθελα απλώς ε, να ευχαριστήσω τους ομιλητές, γιατί είναι πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσει κανείς τι σημαίνει ε, ένα παιδί διαιρεμένο μεταξύ των δύο γονιών μπορεί τελικά να μην γνωρίσει τον ένα από τους δύο γονείς και ήταν και δική μου περίπτωση και επίσης ε, ε, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της, στο ζήτημα της διαμεσολάβησης και ζητώ συγγνώμη και για τη φωνή μου, είμαι άρρωστη. Το πρόβλημα της διαμεσολάβησης ε, ουσιαστικά απευθύνεται το θέμα της διαμεσολάβησης σε ενήλικες γονείς, αλλά πολλές φορές οι γονείς δεν συμπεριφέρονται σαν ενήλικες. Ε, πολλές φορές ε, τα παιδιά είναι το διακύβευμα, είναι όμοιροι και πολλές φορές τα παιδιά φοβούνται να μιλήσουν, να φοβούνται πως φάνε ξύλο κτλ. Εγώ αυτά τα ξέρω απ' έξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ε, πραγματικά εξαιρετικές οι ομιλίες σας. Για μια ακόμη φορά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Μάριο. Κύριος Μαρίνιο Πίντο, θέλει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, την εκτίμησή μου και το θαυμασμό μου για το έργο των ομιλητών. Πολλές φορές είναι μία πολύ δύσκολη δουλειά γιατί δεν ε, υπάρχει κατανόηση από όλους όσους έπρεπε να έχουν ε, λαμβάνει τις ευθύνες τους με διαφορετικό τρόπο. Πριν ε, κάποια χρόνια στην Πορτογαλία ε, ξέρω την υπόθεση ότι η ακρόαση ενός παιδιού από ένα δικαστή ε, κατέληξε στο να ληφθεί μια ορθή απόφαση. Μιλάμε για την περίπτωση ενός διαζυγίου. Ο δικαστής μίλησε στο παιδί, παρουσία όλων και κάποια στιγμή το ρώτησε ποιον καλεί το βράδυ, ποιον φωνάζει το βράδυ όταν φοβάσαι τη μαμά σου ή τον μπαμπά σου ποιον καλείς. Και ήταν καθοριστική η απάντηση του παιδιού για να βοηθήσει το δικαστή να πάρει την απόφασή του. Δηλαδή που υπήρχε ο σύνδεσμος της ιστοργής. Και είναι σημαντικό λοιπόν να ακούσουμε το παιδί. Είναι ένας, ένα ανθρώπινο το παιδί που εκφράζεται και φυσικά όχι όπως ε, οι ενήλικοι με έναν ε, ε, ψευδή και πλαστό τρόπο, αλλά οι ενήλικες θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοήσουν το μήνυμα που θέλει να στείλει το παιδί είτε με τα λόγια, είτε με το βλέμμα, είτε με τις χειρονομίες. Αυτό είναι το κύριο καθήκον ενός δικαστή. Για μια ακόμη φορά, εγώ θέλω δημοσίως να δηλώσω τις ευχαριστίες μου στους ε, ομιλητές μας εδώ και επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, να εκφράσω και τη θλίψη μου για αυτό το θέμα. Στην Επιτροπή αυτή δηλαδή να μην ξυπνά το ενδιαφέρον των συναδέλφων είναι ένα τέτοιο ζήτημα, γιατί δυστυχώς είναι πολύ μικρός ο αριθμός των συναδέλφων που περιβρίσκεται εδώ. Κοιτάξτε, τουλάχιστον έχουμε την παρηγοριά να σκεφτούμε ότι η δουλειά της συναδέλφου μαζί με της κυρίας Αρτιά, μαζί με τον κύριο Τσιεύσκα θα είναι διαθέσιμη σε όλους και θα μπορείτε να τη διαβάσετε γιατί πολύ σπάνιο ο νομοθέτης μπορεί να φτάσει τόσο στην ουσία του ζητήματος όπως κάναμε εμείς σήμερα κυρίες και κύριοι παραθέτοντας πρακτικά παραδείγματα γιατί δεν ε, ε, υπάρχει δυνατότητα να βελτιώσουμε ε, μια κατάσταση όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Και πραγματικά εσείς έχετε τον μπαλάκι στο γήπεδό σας, γιατί εσείς γνωρίζετε τα πράγματα. Έτσι λοιπόν. Εγώ θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό που πήρατε το λόγο και εκφραστήκατε με τον τρόπο αυτό. Θα ήθελα να σου δώσω το λόγο, Ελιζαμπέτ, για τις καταλεκτικές παρατηρήσεις και σε ευχαριστώ για τη δουλειά που έκανες. Ε, από ό,τι φαίνεται, έχει γράψει και 10 σελίδες σημειώσεις, που είναι καλό σημάδι για αυτή, αλλά κακό σημάδι για τη βοηθό της. από ό,τι φαίνεται, ήταν πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη των πάνελ που μας έδωσαν ε, οπτικές, ε, αληθινές, ε, αλλά και αχμηρές για το πώς είναι η πραγματική ζωή των παιδιών αυτών όταν χωρίζουν οι γονείς και μεγενθύνονται τα προβλήματα ε, γιατί έχουμε διασυνοριακά ζευγάρια. Να είστε σίγουροι ότι τα όσα μας είπατε θα αντιτάξουμε στην νομοθεσία και εγώ συντονίστρια για τα δικαιώματα των παιδιών. Θα λάβω υπόψη τα όσα είπατε για να μπορέσω να βελτιώσω τις πολιτικές μας και να ρυθμίσουμε τις υποθέσεις που έχουμε επιτάπητος. Επίσης ε, θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους αλλά και ιδίως εσά, Πρόεδρε και την Επιτροπή Ρομπικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί μας υποστηρίζετε στο έργο μας γιατί υλοποιείτε τέτοιες ακροάσεις ε, και τις βάζετε στο πρόγραμμα της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων αυτό θα σας να προχωρήσουμε, θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε μαζί. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε την καλή δουλειά. Είναι εξαιρετική ομάδα. Και είμαστε ιδιαίτερα κινητοποιημένοι για να σημειώσουμε πρόοδο σε όλα αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Χαίρετε της ευγνωμοσύνης μου. Μάλιστα θα διακόψουμε τη συνεδρίαση για 9 λεπτά λέει ο Πρόεδρος γιατί θα ξεκινήσει μια δεύτερη συνεδρίαση για 45 λεπτά στις 6 παρατέταρτο. Σας ευχαριστώ και πάλι, κυρίες και κύριοι, και έχω την εντύπωση ότι τα όσα μας αναφέρετε σίγουρα θα είναι μέρος των νομοθετικών προτάσεων που θα εκπονήσουμε. Σας ευχαριστώ.